Ja, sehr geehrte Damen und Αγαπητές ε, φίλοι, κυρίες και κύριοι, με την άδειά σας ε, κυρίσω ξανά την έναρξη της ε, απογευματινής πια συνεδριάσεως και συνεχίζεται βεβαίως η συνεδρίαση από το πρωί μετά από εντατικές ακροάσεις που διεξήχθησαν σήμερα το πρωί έχουμε σήμερα το απόγευμα τον Γενικό Διευθυντή της ε, Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχετε αγαπητέ κύριε σήμερα την τιμή να εκπροσωπείτε την ύπατη εκπρόσωπο κυρία Άστον η οποία λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων δεν έσχε την δυνατότητα να είναι παρούσα σήμερα αλλά μας διαβεβαίωσε ότι πολύ ευχαρίστως θα προσερχόταν και βεβαίως εμείς θα θέλαμε να ανταλλάξουμε απόψεις μαζί της, αλλά αντιλαμβανόμαστε και την σημασία των ανηλυμένων της υποχρεώσεων, που αναλαμβάνει βεβαίω κατ' εντολή της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Θα παρακαλέσω πρώτα τα ε, μέλη του ελεκτικού συνεδρίου. Α, ο κύριος, α, μετά ο κύριος Φαζάκας πρώτος, ο κύριος Μουγκουρούζα. Έχετε το λόγο κύριε, ε, μέλος του ελεκτικού συνεδρίου. Κύριε Πρόεδρε και εσείς ε, αγαπητά μέλη, όπως σας είπα το πρωί, το κεφάλαιο 9 της ετήσιας έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναφέρεται στις διοικητικές δαπάνες των θεσμικών και άλλων οργάνων της Ένωσης στο σύνολό τους και δεν ε, προβλέπει αξιολόγηση ανά θεσμικό όργανο. Το κεφάλαιο αυτό ωστόσο περιλαμβάνει συστάσεις που εφαρμόζονται στους διάφορους οργανισμούς και ιδίως βεβαίω εν προκειμένου για την υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Θα σας υπενθυμίσω εν συντομία την προσέγγιση ελέγχου του ελεγκτικού συνεδρίου για το 2012 σχετικά με 151 συναλλαγές που σήμαναν σημαντική αύξηση σε σύγκριση με παλαιότερα χρόνια. Δεύτερο, μια πιο συγκεκριμένη ταξινόμηση των σφαλμάτων στις προμήθειες για να υπάρξει εναρμόνιση σε όλους τους τομείς και να ανταποκρίνονται στα κεφάλαια της εκθέσεως του ελεγκτικού συνεδρίου. Τρίτο, οικονομικό έλεγχο των συστημάτων εποπτείας και ελέγχου των θεσμικών οργάνων. Εν προκειμένου το συνέδριο προβαίνει σε έλεγχο σε βάθος δύο οργάνων τον χρόνο κατά εναλλακτική σειρά. Για το 2012 ήλεγξε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Για το 2013 είναι η Κομισιόν και το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών, ε, της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Και σε ό,τι αφορά την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ελέγξαμε το σύστημα προσλήψεως προσωπικού με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και για τις δηλώσεις αξιοπιστίας για τον έλεγχο του 2015 το ελεγκτικό συνέδριο τότε θα μπορέσει να πει περισσότερα για τα θέματα αυτά. Όπως είπα και σε παλαιότερες παρουσιάσεις, όπως και σε παλαιότερα χρόνια, τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων αυτών είναι θετικά. Και καταλήγει το συνέδριο ότι οι διάφορες συναλλαγές για το 2012 ήταν από κάθε ουσιαστική άποψη εντάξει νομικά και οικονομικά. Και Θεωρεί επίσης ότι τα συστήματα εποπτείας και ελέγχου για τα θεσμικά όργανα, δηλαδή για τις διοικητικές τους δαπάνες, συμμορφούνται με τις απαιτήσει του δημοσιονομικού κανονισμού. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, ίσως να ενθυμίστε ότι στους, ελέγχου ελέγχους του 2011 για την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσεως, το συνέδριο είχε βρει ορισμένα σφάλματα σχετικά με την καταβολή κοινωνικών επιδομάτων και άλλων ευεργετημάτων στα μέλη του προσωπικού, στην διαχείριση ενός, ε, μιας συμβάσεως για την παροχή, συμβάσεων, ε, για την παροχή μάλλον υπηρεσιών ασφαλείας και σχετικά, και άλλα σχετικά. Για το 2012, για τον έλεγχο των λογαριασμών, δεν σημειώθηκε κανένα από αυτά τα σφάλματα σε σχέση με την υπηρεσία εξωτερικής δράσεως, εκτός από περιορισμένα σφάλματα στην καταβολή κοινωνικών επιδομάτων και άλλων ευεργετημάτων για μέλη του προσωπικού. Αυτά τα ελλείμματα οφείλονται και στην έλλειψη ενήμερης πληροφόρησης σε ό,τι αφορά τους φακέλους του προσωπικού που λαμβάνουν επιδόματα και από εθνικές πηγές ή σε ό,τι αφορά την προσωπική τους κατάσταση. Το συνέδριο σημειώνει επίσης ότι οι καταβολές γίνονται από τον Ταμεία της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Και μαζί με, αυτού, με, τα, με, το πρόσωπα, με τα αυτά, το ελεγκτικό συνέδριο ε, τα απαραίτητα μέτρα για, να, για με τις συστάσεις του συνεδρίου. τέλει θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την προσοχή που χαρίσατε στα λόγια μου και ε, να σας διαβεβαιώσω ότι είμαι στη διάθεσή σας για οποιασδήποτε διευκρινήσεις που ενδέχεται να επιθυμείτε. δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Φαζάκας. Ο κύριος Φαζάκας απαντά στα γερμανικά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη. Εύχομαι καλή χρονιά και βεβαίως καλή επιτυχία σε ευρωεκλογέ. Θα τα πω τώρα στα αγγλικά βεβαίως. Μετά από τα όσα είπε ο αξιότιμος συνάδελφός μου, ο κύριος Μουγκουρούζα, για την ε, τακτικότητα και νομιμότητα των συναλλαγών, όπως διαπιστώσαμε, σας ε, πληροφορώ ότι το τρίτο τμήμα του ελεγκτικού συνεδρίου που αναλαμβάνει τον έλεγχο της εξωτερικής ε, δράσης έχει αρχίσει τον οικονομικό έλεγχο των δραστηριοτήτων και βρίσκεται στον αγωγό, βρίσκεται στην τελική φάση πλέον η σχετική έκθεση. Η έγκριση μπορεί να αναμένεται περί τον Μάιο ίσως και τον Απρίλιο. Θα εξαρτηθεί αυτό από την κατατιμωλία διαδικασία αλλά ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να σας υποβάλουμε την έκθεση αυτή πρώτου τέλους της θητείας σας, έτσι ώστε να μπορέσετε, να μπορέσετε να εργαστείτε κι εσείς. Αυτά ήθελα μόνο να σας πληροφορήσω και αναμένω βεβαίως με μεγάλο ενδιαφέρον την περαιτέρω εξέλιξη της διαδικασίας. Ο Πρόεδρος Τόιρερ, ευχαριστώ κύριε Φαζάκας. Έχουμε λοιπόν τώρα τη γνωμοδότηση του ελεγκτικού συνεδρίου και θα παρακαλέσω εσάς Τώρα κύριε Οσάλιβαν να προχωρήσετε στις ε, παρατηρήσεις σας. Thank ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας πω ότι ε, για μένα είναι πραγματικά τιμή και ευχαρίστηση να εκπροσωπώ την ύπατη εκπρόσωπο και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης σήμερα στην Επιτροπή σας και να σας διαβιβάσω το ότι η κυρία Άστον λυπάται ιδιαίτερα, η οποία δεν βρίσκεται σήμερα εδώ πέρα στην Επιτροπή. Ξέρετε ότι ε, έπρεπε να, στη, ταξιδέψει στη Γενέβη για τι ε, διαπραγματεύσει που γίνονται εκεί πέρα για το ζήτημα τη Συρία, αλλά καθώ επίση και για το ζήτημα του Ιράν και πρέπει να κάνει κάποιε δηλώσει και στον ε, τύπο. Ξέρετε, ότι όσοι είδατε σήμερα το πρωί στην τηλεόραση, ήταν στη Γενέβη και Προφανώς δεν είναι δυνατόν για αυτή να βρίσκεται σήμερα εδώ, σήμερα το απόγευμα. Λυπάται πάρα πολύ λοιπόν για την απουσία της. Με την άδειά σας λοιπόν κύριε Πρόεδρε θα ήθελα και να σας διαβάσω αυτά τα οποία θα εκφωνούσε η κυρία Άστο να βρισκόταν εδώ πέρα σήμερα. Αυτές ήταν οι πρώτες παρατηρήσεις που θα κάνω και συνέχεια θα απαντήσω και εγώ σε κάποια ερωτήματα. Οι αρχικές παρατηρήσεις λοιπόν της κυρίας Άστον είναι οι ακόλουθες. Χαίρομαι πάρα πολύ που μου δίνετε για άλλη μια φορά δυνατότητα να αναφερθώ στις δραστηριότητε καθώ επίση και στην εκτέλεση προπολογισμού για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση. Και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι σε θέση να απαντήσω σε ερωτήσει σα. Παράλληλα, περιμένω από εσά κάποιε περαιτέρω ιδέε, γιατί είμαι πεπισμένη ότι θα πρέπει από κοινού να συνεργαστούμε για να καταφέρουμε να χρησιμοποιήσουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο του περιορισμένου οικονομικού πόρου που έχουμε για να καταφέρουμε να ανταποκριθούμε στι προκλήσει που έχουμε τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και στο διεθνέ επίπεδο. Η συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν θεμελιώδου σημασία, ιδίω για του τομεί εκείνου που θέλουμε να προωθήσουμε τι βασικέ αρχέ Ευρωπαϊκή Ένωση. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοδομητική συνεργασία που είχαμε για διάφορου τομεί δράση. Χαίρομαι ιδιαίτερα για την επιτυχία που έχουμε σημειώσει σε διεθνέ επίπεδο, στο διεθνέ προσκήνιο, για τη συμφωνία που έχουμε πετύχει για έναν ε, περαιτέρω διάλογο ανάμεσα στο Κωσυβοπαίδιο και τη Σερβία, για το ότι έχουμε καταφέρει επίση να πετύχουμε πιο στενέ πλέον διπλωματικέ σχέσει ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Ιράν, ιδίω στα πλαίσια των ε, συζητήσεων EU 3 συν 3. Όλες αυτές οι δράσεις συμβάλλουν πάρα πολύ στην παγκόσμια ειρήνη. Καθότι οι προκλήσεις αυτές αυξάνονται και καθότι έχουμε όλο και πιο επικοδομητική συνεργασία, είμαι σίγουρη ότι θα καταφέρουμε να πετύχουμε όλο και περισσότερες επιτυχίες στο μέλλον. Είμαι πεπισμένη ότι θα καταφέρουμε να συνεργαστούμε όλο και περισσότερο με, διεθνούς, με διεθνείς παράγοντες και θα καταφέρουμε να καταλάβουμε κατά αυτόν τον τρόπο την προστιθέμενη αξία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Έχουμε λοιπόν μία αναθεώρηση που γίνεται για την υπηρεσία μου, που προβλέπονται συγκεκριμένε προτάσει και συστάσει για να βελτιωθεί η υπηρεσία αυτή. Ορισμένε έχουν ήδη αρχίσει να εφαρμόζονται, όπω η καλύτερη συνεργασία με τι πρεσβείε στι τρίτε χώρε, καλύτερη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συγκεκριμένη εντολή όσον αφορά του ειδικού εντεταλμένου Ευρωπαϊκή Ένωση. Προβλέπονται επίση μια δεύτερη φάση κάποιε άλλε προτάσει που έχουν να κάνουν με το τέλο του τρέχοντο έτου, του 2014, προκειμένου να έχουμε μια καλύτερη ευθυγράμμιση όλων των διοικητικών δομών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Το 2015 ο νέος ύπατος εκπρόσωπος είναι σε θέση να παρουσιάσει περισσότερες συστάσεις. Δεδομένης της δινης οικονομικη οικονομική κατάσταση, ορισμένα κράτη-μέλη απευθύνονται στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης για περαιτέρω στήριξη, Ιδίως μέσω του δικτύου αντιπροσωπιών που έχουμε παντού στον κόσμο. Η υποστήριξη αυτή βοηθά πραγματικά τι εθνικέ διπλωματικέ αρχές να επικεντρωθούν σε κάποιε εθνικέ εγχώρε προτεραιότητε Έχουμε τακτικές συναντήσει ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική δράση και τα κράτη-μέλη για να πτύξουμε περαιτέρω συνέργειε. Σύμφωνα με το πνεύμα τη συνθήκη τη Λισαβόνα, είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να έχουμε την ενεργό συμμετοχή των κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γι' αυτό το λόγο προτείνουμε και έχουμε προτείνει μέχρι στιγμή σε 14 τρίτες χώρες συγκεκριμένες υπηρεσίες κοινή συνεργασίας. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης βέβαια υπόκειται και αυτή σε συνεχείς δημοσιονομικές πιέσεις. Θέλουμε να κάνουμε σημαντικές βιώσιμες εξοικονομήσεις. Ο προπολογισμός για το 2014 προβλέπει εξοικονομήσεις περίπου 1 εκατομμυρίου ευρώ, ιδίως όσον αφορά τις αποζημιώσεις και τα επιδόματα που δίνονται σε εργαζομένους αντιπροσωπείες και 2,2 εκατομμύρια ευρώ όσον αφορά κυρίως τα ταξιδιωτικά έξοδα των εργαζομένων της Ευρωπαϊκής υπηρεσίε εξωτερική δράσης. Η υπηρεσία μου επίση έχει συγχωνεύσει κάποιες διοικητικές θέσεις, πέντε διοικητικές, μάλλον πέντε διοικητικές θέσεις και εννιά πιο υψηλόβαθμες διοικητικές θέσεις και έχουμε καταφέρει στα πλαίσια του 2013 να πετύχουμε το στόχο μας όσον αφορά την πρόσληψη συμβασιούχων υπαλλήλων σε διοικητικό επίπεδο είναι περίπου το 13% του συνολικού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Έχουμε πολύ σημαντική συνεργασία με τους εθνικούς διπλωμάτες. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ τη συνεργασία που έχουμε με τα κράτη-μέλη. Επίσης, έχουμε προκηρύξει κάποιες θέσεις οι οποίες ήταν ανοιχτές και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η επιτυχία όμως Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης βασίζεται στο να υπάρχουν συνεχή κίνητρα για, τους, για το μόνιμο προσωπικό μας. Ασχολούμεθα λοιπόν με το ζήτημα αυτό και για πρώτη φορά το 2013 αρχίσαμε να χρησιμοποιούμε έναν εσωτερικό μηχανισμό κινητικότητος και έχουμε και έναν νέο εσωτερικό μηχανισμό περιτροπής μετακίνησης των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Μολονότι η κατάσταση δεν είναι ακόμα πλήρω ικανοποιητική, έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδο για να έχουμε καλύτερη εκπροσώπηση των φύλων. Έχει αυξηθεί, διπλασιαστεί μάλιστα από 10 σε 24 ο αριθμό των γυναικών που συμμετέχουν ε, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση, 17% όμω μόνο ακόμα των συνολικών, του συνολικού προσωπικού και έχουμε περίπου 18% συμμετοχή των γενικών, ιδίω όσον αφορά τι ψηλόβαθμε θέσει. Κατά διάρκεια του 2012, πολύ σημαντική πρόοδο επιτεύχθη όσον αφορά την, το διαγωνισμό για τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, όπως είπε και εκπρόσωπος λεκτικού συνεδρίου. Βάσει ενός συγκεκριμένου σχεδίου δράσης έχουμε καταφέρει να καταβάλουμε όλες τις απαραίτητες πληρωμές, έχει μειωθεί το ποσοστό σφάλματος και έχουμε καταφέρει να επεκτείνουμε τις συμβάσεις αυτές σε περισσότερους φορείς. Υπάρχει επίσης μία ad hoc task force για το ζήτημα αυτό, η οποία άρχισε να εργάζεται από τα τέλη του 2013, προκειμένου να έχουμε συγκεκριμένη στήριξη προς τις αντιπροσωπείες ιδίω ιδίως όσον αφορά τη σύναψη ε, συμφωνιών συνεργασίας με ε, εξωτερικούς φορείς στον τομέα παροχής υπηρεσιών ασφάλειας. Ένα άλλο σημαντικό παράγοντα τη επιτυχία Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση είναι ότι έχουμε καταφέρει να έχουμε μια αμοιβαία επικοδομητική συνεργασία με όλα τα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αρχής γενομένη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθώς επίσης όμως και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπου είμαι αντιπρόεδρος υπεύθυνη για ζητήματα συνοχής εξωτερικής δράσης και υποστηρίζομαι την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του Service Level Agreement, τη Συμφωνία Επιπέδου Εξυπηρέτηση. Πολύ καλή συνεργασία έχουμε επίση και με το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο και χαίρομαι πάρα πολύ που τα μέλη του βρίσκονται εδώ πέρα σήμερα καταφέρνουμε να προωθήσουμε συγκεκριμένα προγράμματα εξωτερικής δράσης. Έχουμε επίσης προγράμματα ελέγχου των, της εξωτερικής μας δράσης, αναφέρθηκε ο κύριος Φαζάκας αυτό, και προσβλέπουμε να έχουμε τους επόμενους μήνες περαιτέρω συστάσεις από το λεκτικό συνέδριο για να βελτιώσουμε τη λειτουργία μας. Συνεργαζόμαστε όμως και με την Όλαφ προκειμένου να καταφέρουμε να επιλύσουμε κάποια προβλήματα που έχουν προκύψει και προκειμένου να ενισχύσουμε όλη τη δράση κατά της ΕΠΑΤΗΣ στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Υπάρχει μάλιστα ένα μνημόνιο κατανόησης με την Όλαφ το οποίο ελπίζουμε ότι θα ολοκληρωθεί και θα συνεχθεί το συντομότερο δυνατό. Συντονίζουμε επίσης τις δραστηριότητές μας με τη Γενική Γραμματεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκειμένου να έχουμε μια συνεκτική δράση πανευρωπαϊκά. Η δράση αυτή συντονισμού απέτησε λίγο παραπάνω χρόνο από ό,τι περιμέναμε, αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε σε θέση πολύ σύντομα να υπογράψουμε αυτή τη συμφωνία, το μνημόνιο μάλλον κατανόησης, τις επόμενες εβδομάδες ή μέρες. Εν κατακλείδη να σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης έχει πλέον παγιώσει τη θέση της στο διεθνές προσκήνιο. Ωστόσο, παραμένουν διάφοροι τομείς όπου η υπηρεσία μου εργάζεται ακόμα προκειμένου να καταφέρει να παγιώσει τη θέση της. Στην ετήσια έκθεσή μας βλέπουμε ότι θέλουμε να έχουμε μια καλύτερη διαχείριση του ετήσιου προπολογισμού μα. Βλέπουμε ότι το ποσοστό σφάλματος ήταν πολύ χαμηλό. Το 2012 το ουσιαστικό σφάλμα ήταν 0,51% στην αφορά τις αντιπροσωπείε και 0,69% στην αφορά την έδρα τη Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση. Και όπω είπε σήμερα, το λεκτικό συνέδριο δεν έχει εντοπίσει σημαντικέ αδυναμίε στου τομεί εκείνου που έκανε έλεγχο και του οποίου αναφέρει στην ετήσια έκθεσή του. Οι απαντήσεις που έχουμε δώσει ελπίζουμε ότι καταδεικνύουν το ότι θέλουμε να έχουμε ένα στο επίπεδο διαφάνειας και ελπίζουμε ότι σας καλύπτουν. Προσβλέπω στη συνέχιση της συζήτησης αυτής και της επικοδομητικής συνεργασίας που είχαμε μέχρι σήμερα. Αυτή είναι η δήλωση που θα έκανε η πατή εκπρόσωπος κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε κύριε Σάλιβαν. Τώρα μπορεί να ξεκινήσει η συζήτηση με τα μέλη της Επιτροπής μας και δίνω καταρχάς το λόγο στον κύριο Ντάμας Ντόιτς, ο οποίος είναι ο συγητής μας.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 Ευχαριστώ. Τώρα σας ακούμε. Θα ήθελα πρώτα να απευθύνω το καλό ορίσατε σε όλα τα προσκεκλημένα μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των άλλων υπηρεσιών πριν να κάνω ορισμένε ερωτήσεις. Όπως γνωρίζετε, η υπηρεσία εξωτερικών δράσεων είναι πολύ νοπή μόλις από το 2011 δρά ανεξάρτητα και το ίδιο αυτό έτος, ή μάλλον αμέσως μετά, το 2012, η Υπηρεσία Εξωτερικών Δράσεων προσέλαβε συνεργάτες συνολικά Πολλού 6.800. Ο προπολογισμό του οργάνου είναι το ένα θέμα. Υπάρχουν βεβαίω και υπάρχει ένα μέρος του προσωπικού που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το 2010 αν έρχεται σε 757.000 ευρώ, χρήμα των φορολογουμένων εννοείται. Σας συνάντησα και σας προσωπικά κύριε Γενική Διευθυντά και ήταν πραγματικά καρποφόρα η συνεδρίαση. Θυμώ να σας ευχαριστήσω τώρα και βεβαίως σας ευχαριστώ κιόλας για το γεγονός ότι απαντήσατε γραπτός στο ερωτηματολόγιο που σας υποβάλαμε με συνολικά 37 ερωτήσεις. Αυτές ακόμη δεν έχουν αναλυθεί. Βεβαίω ήταν βραχύτατη η προθεσμία, δεν ευθύνεται όμως η γραμματεία γι' αυτό. Σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση των απαντήσεων, έχω εδώ να μπορώ να διακρίνω τρεις ομάδε. ομάδες ανάλογα με την σημασία τους. Πρώτα, το προσωπικό ή το εισόδημα του προσωπικού, μετά το διαχειριστικό κόστος. Αρχίζω τώρα με αυτά που περιλάμβανε η έκθεση του 2011. Πρόκειται για υπηρεσία η οποία έχει υψηλό κόστος. Αυτό το λένε οι εμπειρογνώμονες. Υπερβολικά υψηλό κόστος. Εάν πρόκειται για κατασπατάληση πόρων ή όχι, αυτό δεν το γνωρίζω, ούτε πρόκειται να το ξεκαθαρίσω. Πρόκειται πάντως για, τις, για διπλωματικές εκπροσωπήσεις που έχουν το υψηλότερο κόστος στον κόσμο. Η, ο αριθμός των συνεργατών με βαθμό AD είναι 510 και από αυτούς ένα μεγάλος αριθμός είναι AD 12 πάει να πει ότι είναι σε πολύ ψηλέ θέσεις είναι λοιπόν εμπροστοβαρής κατά κάποιο τρόπο ο οργανισμός δηλαδή σημαίνει ότι το βάρος συγκεντρώνεται ψηλά πώς είναι δυνατόν πώς εξηγείται ότι υπάρχουν τόσο υψηλόβαθμα στελέχη άντε 12 και παραπάνω και αυτό σημαίνει δαπάνες της τάξη των 500 των, συγγνώμη, των 5 εκατομμυρίων ευρώ τον μήνα. Και αν συνυπολογιστούν και οι δαπάνες για τους συνεργάτες των αντιπροσωπιών, δηλαδή διάφορα επιδόματα και πέραν των καθαρών απολαβών τους, τότε το ποσό βεβαίως ανέρχεται. Αυτά αφορούν τους συνεργάτες των αντιπροσωπιών. Και σε νούμερα απόλυτα αυτό σημαίνει άλλα περίπου 5 εκατομμύρια το μήνα. Συνολικά δηλαδή 10 εκατομμύρια ευρώ το μήνα. Κύριε Γενική Διευθυντά, που, σε τι οφείλεται ότι το ποσοστό των υψηλόμισθων είναι πάνω από 15%. Ξαναλέω, υπάρχουν πολύ υψηλόμιστοι συνεργάτες σας. Το θεωρείτε δικαιολογημένο αυτό, να μιλούμε για τέτοια ποσά. Σε ό,τι αφορά τώρα τις συντάξεις για το 2012 ή 2013, συνταξιοδοτήθηκαν 109 συνεργάτες σας και ο μέσος όρος των συντάξεών τους ήταν της τάξης των 5.800 ευρώ. Υπάρχουν συνταξιοδοτούμενοι μεταξύ αυτών, των οποίων συντάξεις ανέρχονται στις 10.000 και πλέον ευρώ. Και υπάρχουν και άλλοι πολλοί οι οποίοι βρίσκονται σχεδόν στο όριο της συνταξιοδοτήσεως. Έχετε κάποια στρατηγική για να χρηματοδοτήσετε τις συντάξεις αυτές. Διότι υπάρχουν εδώ υποχρεώσεις καταβολής συντάξεων που οφείλετε να τηρήσετε. Η τρίτη μου ερώτηση αναφέρεται στα επιδόματα κατοικίας για το 2012 στις αντιπροσωπείες έχετε 675 συνεργάτες που λαμβάνουν ή έλαβαν επίδομα κατοικίας της τάξης συνολικά των 30 εκατομμυρίων ευρώ. Δηλαδή, ανα μήνα και ανακεφαλή περίπου 3.700 ευρώ. Τέτοια ποσά έλαβαν ως επίδομα κατοικίας οι ε, συνεργάτες σας αυτοί. Από το 2014 θα ασκηθεί νέα πολιτική, θα υπάρξει δηλαδή μια οροφή, ένα ανώτατο ποσό, Δεν υπάρχει επομένω άμεση διασύνδεση με το 2012, γιατί όπω είπα η νέα ρύθμιση θα αρχίσει να ισχύει από το 2014. Αναρωτιέμαι όμω πώ αποφασίστηκε αυτή η οροφή. Από τις 140 αντιπροσωπείες, αυτή εισάγεται σε 89. Παραμένω πάντα στο κόστος του προσωπικού. Μετά το 2012 άρχισε να ισχύει ένας κανονισμός προσωπικού, staff regulation, η οποία επιτρέπει, ο οποίος μάλλον επιτρέπει ήδη εξοικονόμηση 2 εκατομμυρίων ευρώ. Η ύπατη εκπρόσωπος το αναφέρει αυτό στην επιστολή της και αυτή προέρχεται κυρίως από την μείωση των επιδομάτων των συνεργατών των αντιπροσωπιών. Εσείς δηλαδή επιβάλλετε μια οροφή για τα επιδόματα κατοικίας, εξορθολογίζεται ακόμη περισσότερο τι δαπάνε προσωπικού. Ποιε εξοικονομήσει αναμένεται από αυτά τα μέτρα. Τέλος, ο τοπικός εργαζόμενος, ο local agent, την η επόμενη ερώτησή μου. Το 2012 είχατε 3.160 τοπικούς εργαζόμενους στις υπηρεσίες της ε, υπηρεσίας εξωτερικής δράσεως. στους οποίους κατεβλήθησαν 160 εκατομμύρια ευρώ που σημαίνει άνω των 3.000 ευρώ ανα κεφαλή και ανα μήνα. Δεν είναι και κανένα σήμα το ποσόν σε σύγκριση με τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Δεν μου φαίνεται δηλαδή να είναι κάπως συγκρίσιμος με τον ελάχιστο μισθό στην Ευρώπη. Η ερώτησή μου λοιπόν τώρα έχει ως εξής. Επί της 100. Πώς επιλέγονται μάλλον τα πρόσωπα αυτά, πώς είναι local agents και ποια είναι τα κριτήρια για τον υπολογισμό των απολαβών τους. Δεύτερο, Αναφέρομαι στους ειδικού απεσταλμένους. 11 τον αριθμό. Συν 100 άτομα βοηθητικό προσωπικό. 11 δηλαδή ειδικοί απεσταλμένοι συν το βοηθητικό τους προσωπικό 30 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Κατά την ίδρυση της Υπηρεσίας Εξωτερικών Δράσεων υπήρχε η πρόθεση να εξορθολογιστεί το σύστημα αυτό των ε, ειδικών απεσταλμένων. Το σύστημα ωστόσο παρέμεινε, ως είχε. Ερώτηση λοιπόν, γιατί δημιουργήθηκε η υπηρεσία εξωτερικής δράσεως και τέθηκε βέβαια το ερώτημα εάν μπορεί να λειτουργήσει, μπορεί να αποδώσει το σύστημα των ειδικών απεσταλμένων, βλέπω όμως ότι παρέμεινος είχε. Πώς μπορεί όμως να μετρηθεί η αποδοσή τους. Η πλειονότητα των ειδικών απεσταλμένων εργάζονται για την λύση κρίσεων, για την επίλυση κρίσεων. Τα καθήκοντά των βεβαίως είναι ειδικά, αλλά οι περισσότεροι από αυτούς διαθέτουν συμβάσεις αορίστου χρόνου, παρόλο που καλούνται να λύσουν συγκεκριμένα προβλήματα. Εργάζονται όμως επί έτη και έτη. Πώς μετράτε εσείς την αποδοτικότητα της εργασίας τους. Πρώτο τελευταίο θέμα, συμβάσεις ασφαλείας. Θέμα το οποίο τέθηκε ήδη και για την έκθεση του 2011 ο Διευθυντής κ. Σάλιβαν είχε ήδη εκφράσει κάποιες επιφυλάξεις σχετικά με τις συμβάσεις με τη Λιβύη ειδικότερα και το Αφγανιστάν που ενέκειτο το πρόβλημα με τις συμβάσεις αυτές. Η υπηρεσία εξωτερικής δράσης είχε φτιάξει ένα σχέδιο για το 2011. Γιατί όμως εσείς έχετε εκφράσει επιφυλάξεις. Άλλο, ερωτικό, άλλο σημαντικό θέμα, ερώτημα. Στην τελική εκτίση έκθεση του το 2011 δηλώνει η υπηρεσία εξωτερικής δράσης ή τουλάχιστον υπόσχεται ότι πρόκειται να συνάψει, να συνυπογράψει μνημόνιο συνεννόησης με την Όλαφ. Τελικά αυτό δεν έγινε. Γιατί δεν συνήθει αυτό το Memorandum of Understanding. Η Όλαφ εξέτασε το 2011 52 υποθέσεις όπου ενεπλέκετο και η Υπηρεσία Εξωτερικών Δράσεων. Και τέλος, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, άλλο σημαντικό οικονομικό θέμα στην τελική έκθεση δραστηριοτήτων της υπηρεσίας το 2012 αναφέρεται ένα ποσό 6,5 εκατομμυρίων ευρώ που εκκρεμούν. Βρίσκονταν λοιπόν σε λογαριασμό της υπηρεσίας αυτά τα 6,7 εκατομμύρια ευρώ έχουν τώρα αυξηθεί, έχουν γίνει 9,9. ...50.000 μονομένες υποθέσεις. Αλλά ποια είναι η εξήγηση. Χρειάζεται κάποιο σχέδιο διαχείρισης εκ μέρους σας, το οποίο να ε, βοηθήσει την επίλυση των ε, εκκρεμών αυτών υποθέσεων. Να επαναλάβω το τελευταίο σημείο, λες ελληνικά. Στα αγγλικά. Ξανά αγγλικά. Ο κύριος Ντόιτς συνεχίζει. Υπάρχουν θέσεις στο λογαριασμό του 2012 6,7 εκατομμυρίων ευρώ. 46.000 ανοιχτές θέσεις και υπάρχουν και άλλα ποσά τα οποία εκκρεμούν. Τα οποία έχουν αυξηθεί από 6,7 εκατομμύρια και έχουν ανέλθει στο ποσό των 8,9 εκατομμυρίων, λέει τώρα ο κ. Στόιτς. Δηλαδή συναλλαγές οι οποίες άρχισαν αλλά εκκρεμούν, δεν έχουν ολοκληρωθεί. Πού οφείλεται αυτό, ότι υπάρχουν ακόμα τόσες εκρεμίσεις πληρώμες. Ευχαριστώ για τη συνεργασία και ελπίζω να μπορέσετε να απαντήσετε. Ευχαριστώ. δέσμοι ολόκληρη ερωτήσεων του εισηγητού για λόγους οικονομίας χρόνου προτείνω να ακούσουμε και τις άλλες παρεμβάσεις αν υπήρχε ε, δυνατότητα δύο ε, πρόσληψη προσώπων από δύο έδρες, τότε θα είχαμε ίσως και μεγαλύτερα, μεγαλύτερες εξοικονομήσεις. Κύριε Πρόεδρε, είμαι σκιώδης εισηγητής και δεν μπορώ να πιστεύω στις λεπτομέρειες. Γιατί θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με την ειδική έκθεση του Ελληνικού Συνεδρίου που μιλάει για την πλησματική χρήση των κοινωνικών πόρων. Όπως είπε ο εισηγητής, πρόκειται για μια νέα υπηρεσία που συγκροτήθηκε, οπότε έχουμε τώρα τα, τις βασικές αρχές που εφαρμόζουν. Πρέπει να πηγαίνουν παντού οι διπλωμάτες υπηρεσίας αυτής, άρα τα πράγματα είναι περίπλοκα. Οπότε και έχουμε το θέμα του να έχουν τις πληροφορίες, υπάρχουν ε, καθυστερήσεις και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη Τότε κατά τη διάρκεια του οικονομικού ελέγχου δεν είχαμε ε, διαπίστωση κάποιων προβλημάτων, κάτι σε σχέση με τα κοινωνικά επιδόματα είχε επισημανθεί, αλλά ό,τι πρόβλημα επισημάνθηκε επελήφθη. το 2012 είχε πάρα πολύ χαμηλό ποσοστό δαπανών διοικητικών κάτω από 2% ήταν το ποσοστό του σφάλματος σύμφωνα με τη διαπίστωση του ελληνικού συνεδρίου. Πέρσι όταν τα συζητήσαμε, ότι θέλουμε να υπάρχει καλύτερη κατανομή, αναχώρα και αναφύλλο. όσον αφορά το προσωπικό, ε, που φυσικά προέρχεται από τις Εθνικές μοντικές Υπηρεσίες. Βέβαια, έχει σημειωθεί πρόοδος. Και επίσης τα πράγματα πάνε καλύτερα όσον αφορά τα, τις υπηρεσίες ασφαλείας σε ε, χώρες ε, όπου υπάρχει κίνδυνος Επίσης βελτιώθηκε η συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, την οποία και ευχαριστώ για τις άκρως ικανοποιητικές απαντήσεις που παρέσχουν στις ερωτήσεις που υποβάλαμε. Κυρία ευχαριστώ. Ακούω παράπονα και από ε, συναδέλφους της επιτροπή Εξωτερικών. Τέλος πάντων, ε, χαίρομαι που ο κ. και είναι παρόν. Σας συγχαίρω κιόλα που ε, τοποθετήσετε τώρα στο γραφείο του Σουάσιγκτον. Αλλά γιατί εκπίπτει η θέση σας, είναι περιττή. Μπορείτε να εξηγήσετε κάπως. Μετά αυτό που εξήγησε ο Τάμας Ντόιτς των ειδικών αντιπροσώπων οι απεσταλμένων. Εκεί εμείς έχουμε ξεσηκωθεί πραγματικά. Προσπαθήσαμε ήδη στην διάρκεια των συζητήσεων για τον προϋπολογισμό με το Συμβούλιο να ενταχθούν δηλαδή οι ειδικοί απεσταλμένοι στην υπηρεσία εξωτερικών δράσεων. Για το 2011 έως 2013 έχουμε αύξηση κόστους των 12 αυτών προσώπων κατά 70%. 70%. Πώς δικαιολογείται αυτή η αύξηση και ούτε καν περιλαμβάνονται οι δαπάνες ταξιδιών τους που έχουν τριπλασιαστεί. Τότε προτείνω να αφήσουμε αυτούς 12 να κάνουν ό,τι κάνουν και να καταργήσουμε την υπηρεσία εξωτερικών. Ακούμε και την πρόταση να δοθεί διοικητική υποστήριξη από την υπηρεσία εξωτερικών στου 12 αυτού απεσταλμένου, αυτό τι σημαίνει, ότι δεν θα έχουμε πλέον καμία επισκόπηση πάνω, καμία εποπτεία πάνω στον προπολογισμό τη υπηρεσίας εξωτερικών δράσεων. Προσοχή λοιπόν. Εδώ θα χυθεί αίμα, μεταφορικά το λέω βέβαια. Ε. Είμαστε, όπω είπα, επιποδός πολέμου. Επίσης, εσείς έχετε προβάλει επιφύλαξη για θέματα συμβάσεων ασφάλειας και ειδικά για την εταιρεία Arbus Security στην Κύπρο. Η Arbus έλαβε από την Υπηρεσία Εξωτερικών Δράσεων τόκους 5.900 ευρώ για καθυστέρηση επί 60 ημέρες 33.000 ευρώ, καταβολή 33.000 ευρώ. Πρόκειται για μια εταιρεία για τη συμβάση της οποίας προφανώς έχετε επιφυλάξεις. Πώς είναι δυνατόν να λάβει η εταιρεία αυτή 5.500 ευρώ για μια καθυστέρηση λίγων χιλιάδων ευρώ. Δηλαδή μήπως μπορώ να καταθέσω χρήματα σε εσά για να αυξάνονται. Παρόμοιες υποθέσεις με την British Telecom. Πάλι με τόκους υπερημερίας. Ε, πρόκειται, εδώ πρόκειται για πραγματική τοκογλυφία. Μήπως μπορείτε να μας εξηγήσετε. Εδώ και χρόνια εγώ ανησυχώ επίσης για την γεωγραφική εξισορρόπηση των συνεργατών και μάνατζερ της υπηρεσίας των εξωτερικών υποθέσεων. Βλέπω τώρα ότι το Συμβούλιο αλλά και τα πρόσωπα που αναφέρετε εσείς ως stock manager στην ιστοσελίδα για το 2011 ήταν 17 ε, θέσεις για το 2013 18 τέσσερις από το Ενωμένο Βασίλειο, τώρα πέντε από το Ενωμένο Βασίλειο. Το 2011 είχαμε τρεις Γάλλους, δύο Ολλανδούς και δύο Σουηδούς, τώρα έχουμε πέντε από το Ενωμένο Βασίλειο, μετά τρεις ε, Γάλλους, τρεις Γερμανούς και έναν από τους υπολείπους. Καμία σχέση με οποιαδήποτε γεωγραφική καταμέριση. Φαίνεται πολύ καθαρά ότι έχουμε σαφέστατη κυριαρχία των Βρετανών στην υπηρεσία αυτή. Τώρα να δούμε και τους heads of delegation, οι διορισμοί που έχει κάνει η κυρία Ήπατη εκπρόσωπος για το 2010 έως 2013, έχουμε διορισμούς 15 Γάλλους, 14 Ισπανούς, 9 Γερμανούς, 9 Ιταλούς, 9 Ουκρανούς και 9 ε, Βέλγους. Πάλι εκεί έχετε διαλέξει τους καλύτερους ή απλά πρέπει κανείς να επιμένει έτσι ώστε τελικά να διοριστεί. Όμως μπορείτε να πείτε κάτι και εδώ. Και μετά θα θέλαμε και κάποια στατιστικά δεδομένα τα οποία αφενός να είναι αξιόπιστα και αφετέρου συγκρίσιμα. Ευχαριστώ. Ο πρόεδρος Τόιρερ. Ευχαριστώ κυρία Κρέσλε. Ο κύριος Γιάν Μιούλντερ. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Να συγχαρώ τον κύριο Σάλιβαν και τον ε, διορισμό του αυτό, ενδεχομένως στην Ουάσιγκτον. Μία ερώτηση για την οποία δεν δόθηκε απάντηση στα έγγραφα τα οποία μας απεστάλησαν. Προτού δημιουργηθεί η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, λέγαμε ότι τα κράτη-μέλη θα εκμεταλλεύονταν την ευκαιρία για να δημιουργήσουν ή να συγκεντρώσουν τις προξενικές υπηρεσίες στα ίδια κτίρια τα οποία αυτή τη στιγμή καταλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Και κατά αυτόν τον τρόπο θα γινόταν μια κάποια εξοικονόμηση πόρων και θα ήταν ε, πολύ πιο εύκολο και τους πολίτες να γνωρίζουν ε, από πού μπορούν να πάρουν βίζα για παράδειγμα για μια ευρωπαϊκή χώρα. Τι γίνεται λοιπόν με την αρχική αυτή ιδέα. Είναι μια ιδέα για την οποία θα δοθεί μια συνέχεια, θα ελοποιηθεί ή όχι. Σας ευχαριστούμε κύριε Μούλντερ. Ο κύριος Σαλαφράγκα έχει το λόγο. Πλήρες μέλος, ε, τακτικό μέλος δηλαδή της Επιτροπής Εξωτερικών. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε ο Σάλιβαν. Πέρσι, εγώ ήμουν συγκριτή της ε, ΑΦΕΤ για την απαλλαγή του 2012 και η έκθεση την οποία παραδώσαμε στην ε, έκθεση δημοσιονομικού ελέγχου είχε την εξήγηση του τι έγινε στην πρώτη σας ε, χρονιά όπου τα πράγματα για πρώτη χρονιά πήγαν καλά. Σήμερα άκουσα την εισήγηση του ε, εισηγητού του Ελληνικού Συνεδρίου. Τα πράγματα δεν μπορεί να είναι τέλεια, αλλά έχετε επιφέρει κάποιες βελτιώσεις. Αναγνωρίζουμε τι προσπάθειές σας. Ε, πρόκειται για μια νέα υπηρεσία, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και θυμάμαι, ήμουν εδώ, όταν ήρθε η Λίδια να μας εξηγήσει τις προσπάθειες οι οποίες κατεβλήθησαν στην αρχή. Άκουσα ότι είπε ο συνάδελφος που έκανε την εισήγηση ότι πρόκειται για την πιο ακριβή υπηρεσία. Αυτό δεν με προβληματίζει γιατί νομίζω ότι θα πρέπει ο πύχης ο δημοσιονομικός να βρίσκεται στο ύψος το οποίο θέλουμε να βρίσκεται η πολιτική μας. Θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί και να μπορούμε να δράσουμε στο πλαίσιο το οποίο τάσεται από τις δημοσιογικές προοπτικές και από τις συνθήκες. Με προσοχή, κύριε Σάλιβαν, μελέτησα αυτό το ερωτηματολόγιο, το εκτενές και νομίζω ότι αυτό το οποίο προέκυψε είναι ότι οι δραστηριότητες σας διέπονται από διαφάνεια. Όχι εισηγητής σε κάποια ερώτηση όσον αφορά τις συντάξεις. Με προσοχή εγώ διάβασα τι έλεγε αυτό το ε, ερωτηματολόγιο και έχουμε δέσει τις συντάξεις των 10.000 ε, συντάξεων και άλλες οι οποίες βρίσκονται στα χίλια κάτι ευρώ. Πρέπει να δούμε πού θα είναι η... ο μέσος όρος να είναι κάτι δηλαδή το οποίο να αντιστοιχεί με το καταστατικό γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι η υψίστη σύνταξη η μεγίστη μετά από 30 χρόνια για κάποιον υπάλληλο είναι το 70% του τελευταίου μισθού. Οπότε θα πρέπει ε, να μην θεωρήσουμε ότι υπάρχει διαφορά ανακατηγορία, αλλά θα πρέπει να δούμε το πώς το σύστημα των συντάξεων θα είναι βιώσιμο. Γιατί όπως ε, είπε και ο συγκητής, έχουμε πάρα πολλούς υπαλλήλους σε διάφορους βαθμούς που τελικά καταλήγουν να εισπράξουν με πολύ μεγάλες συντάξεις. Είναι ε, κάτι το θετικό, η διαδικασία πρόσληψης των επικεφαλής των ε, ε, αντιπροσωπιών των, και οι υπουργοί ορίζουν τους πρέσβεις και υπάρχουν κάποια πάνελ τα οποία λειτουργούν. Επομένως, με το δεξί ξεκίνησε η υπηρεσία, έχει κινητικότητα, έχουμε αυτό το επιτυχέ οδηματολόγιο και άρα θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε ως κριτήρια ε, τα προσόντα και τι ικανότητε για τις προσλήψεις. Θέλω να σταθώ σε τρία σημεία. Πρώτα απ' όλα θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να προχωρήσουμε όσο μπορούμε καλύτερα στο να συναυθεί η σχετική συμφωνία με την Όλαφ. Πρόκειται για μια υπηρεσία που θα πρέπει να περιβάλλεται από κάποιες εγγύσεις. Και θα πρέπει να έχετε καλές σχέσεις και στην καλή συνεργασία με την Όλαφ. Όμως υπάρχει κάτι κύριε Σάλιβαν, το οποίο ίσως δεν είναι στενά αρμοδιότητά σας το Κοινοβούλιο ενεργά είχε αναμειχθεί στα πλαίσια της συναπόφασης για την έγκριση των διαφόρων ε, ε, οικονομικών εργαλείων. Πριν πάντως ολοκληρωθεί η αναπτυξιακή ενίσχυση και χρηματοδότηση, είχαμε αποσύρει 80 υπαλλήλους από τις αντιπροσωπείες θεωρώντας ότι η πρόταση της Επιτροπής θα κατήσχε. Όμως δεν ίσχυσε κάτι τέτοιο, δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Κάποιες χώρες βγήκαν από τη συνεργασία, μετά ξαναμπήκανε στα πλαίσια της συναπόφασης. Έτσι αποφάσισε Συμβούλιο και η Επιτροπή. Οπότε, τελικά, ήταν λάθος το να προδικάσει κανείς το αποτέλεσμα της ε, διαπραγμάτευσης. η ΑΦΕΤ σας ζήτησε το τι θα γίνει και η Επιτροπή Ελέγχου σας το ζήτησε. Ανοίξατε τρία, τρεις υπηρεσίες στο Σουδάν, στη Λιβύη, στη Μιανμάρ και τα τρία δικαιολογούνται λόγω των πολιτικών που ασκούμε. Αλλά θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο ρόλος του Παναμά μετά από τη Συμφωνία Σύνδεση έχει καινούριο ρόλο και έχουμε τώρα σχέση με αυτή τη χώρα. Θα πρέπει να έχουμε την αντιπροσώπευση που αντιστοιχεί στο επίπεδο των σχέσεών μας και της σημασίας αυτών. Το ξαναζήτησε φέτος αυτό η ΑΦΕΤ. Νομίζω ότι το μελετάτε εσείς και σας παρακαλώ αν μπορείτε πέστε μας δύο λόγια όσον αφορά το ζήτημα αυτό. Τελευταία ερώτηση και κλείνω κύριε Πρόεδρε. Εργάζομαι στην Επιτροπή που ασχολείται με τα της Αμερικανικής Υπηρεσίας Ασφαλείας. Όπως ξέρετε έχουν στοχεύσει και εμάς αυτές οι υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ. Για πέστε μου, αναβαθμίσαμε την ασφάλεια των αντιπροσωπιών μας επί τη βάση αυτών των νέων. Ισχύει λοιπόν τέτοια αναβαθμισμένη ασφάλεια των υπηρεσιών μας στη ΣΥΠΑ και στην Ουάσιγκτον συγκεκριμένα. Ευχαριστώ πολύ λέει ο Πρόεδρος. Έχουμε αυτή τη δεσμή ερωτήσεων και περιμένω πώς και πώς και ψάχνω να ακούσω τις απαντήσεις σας. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους αξιότιμους βουλευτάς για τις παρατηρήσεις τους, τις ερωτήσεις, τις οποίες θα προσπαθήσω να απαντήσω. Βέβαια, αν απαντήσω σε όλους, θα σας φάω όλο το χρόνο, δεν θα το κάνω Γι' αυτό που είπε ο ο κ. Ντόιτσο. 500 εκατομμύρια είναι η προοικοδότησή μας, δεν ξέρω αν είναι πιο ακριβή υπηρεσία, γιατί έχουμε τους υπαλλήλου που πληρώνονται σύμφωνα με το καταστατικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσο περίπου αναλώνει το βελγικό υπέξ, το οποίο βρίσκεται κάπου στον ευρωπαϊκό όρο Γιατί στα μεγάλα ευρωπαϊκά κράτη τα υπέξ έχουν προπολογισμούς πολλαπλάσιους. Άρα, ούτε είμαστε ακριβοί, ούτε φθηνοί. Έχουμε αυτές τις 49 πόσες έχουν αντιπροσωπείες και τελικά το κόστος δεν καθορίζεται από εμά, καθορίζεται από εσά. Βάσει των όσων τάσει ο νόμος, για την αμοιβή των υπαλλήλων μονίμων ή προσωρινών. Όσον αφορά τις συντάξεις ισχύει το ίδιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενταξεις ισχυει το συνταξιδοτικό αυτό το συνταξιδοτικο αυτο ταμειο και αυτό ισχύει για όλα τα θεσμικά όργανα. Επί τη βάση του καταστατικού. Εγώ υπηρετώ πάρα πολλά χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το αν είναι υψηλέ συντάξει αυτό τελικά είναι πολιτική χρήση, αλλά τελικά υπάρχει αυτή η αυτοχρηματοδότηση. Τα δέκρατη μελη σύμφωνα αυτό το σύστημα, πλήρωναν αυτό το ταμείο, αλλά ποτέ σε εμά δεν έπρεπε να εισφέρουν. Άρα τελικά νομίζω ότι οι συντάξεις δεν έχουν κοστίσει και πολλά στα κράτη-μέλη. Βεβαίω και μπορεί κανεί να συζητήσει τα, το, το κατά πόσο πληρώνονται πολύ ή λίγο με τους μισθού οι ευρωεπάλληλοι. Αλλά όσον αφορά το στεξιδοτικό, αυτό είναι άσχετο παντελώ με μας. Όμως, Υπάρχει εντάξει, κάποιος ε, ψηλόδρομος υπάλληλο μπορεί να παίρνει ψηλό μισθό. Είναι μια περίπτωση, έτσι υπολογίζεται. Όσον αφορά τώρα την πυραμίδα του προσωπικού, κύριε Ντόιτσο, κάτι το οποίο αποτελεί πάγιο θέμα συζήτηση. θέλω απλώς να σας πω δύο πράγματα. Έχουμε θέμα δημογραφικό. Ξέρετε ότι όταν κάποιοι υπηρετούν επί μακρόν, στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτομάτως προωθούνται στην πυραμίδα. Και όπως πέραν τα χρόνια ξεκινούν AD5 και μετά καταλήγουν AD12 εάν έχουν εργαστεί όπως πρέπει κλπ. Άρα αυτό το οποίο μπορεί να πει για την εξωτερική υπηρεσία είναι ότι είναι μια υπηρεσία γυράσκουσα, όχι παλαιά, γυράσκουσα. Γιατί κληρονομήσαμε από την Κομισιόν και από το Συμβούλιο προσωπικό που βρίσκεται στο ας πούμε δεύτερο μήχρονο, στο δεύτερο ήμιση της σταδιοδρομίας τους και η μέση μας ηλικία είναι περί τα 45 αν όχι πιο κοντά στα 50. Οπότε το θέμα το οποίο έχει συζητηθεί στο παρελθόν και το είπαμε και με την κυρία Γκρέσλε είναι ότι και από τα κράτη-μέλη προσλάβαμε προσωρινούς οι οποίοι είναι ήδη υψηλόβαθμοι και έπρεπε να υπηρετήσουν σε θέσεις ευθύνης αντιπροσωπείας. Σας βεβαιώ ότι επίσης ε, προσλάβαμε και με βαθμό AD5, AD7 και γι' αυτό κατηγορηθήκαμε όμως και θυμάμαι ότι είχε πει η Λεβιάστον ότι να σας ξαναπώ έχω εδώ τα στοιχεία. Τα είπαμε, δεν πούμε. Από AD 15 16 πήγαμε στο AD 6 και 7. Δηλαδή αλλάξαμε τελικά τη μορφή της πυραμίδας. Αλλά τελικά όλα είναι θέμα ηλικία των υπαλλήλων. Τώρα φορά αφορά τις δαπάνες ε, φιλοξενίας, στέγασης, Πάλι θεωρούμε ότι και επ' αυτού ότι είμαστε στο μέσο όρο. Οι πρεσβευτές μας μένουν σε ακίνητα τα οποία πάλι βρίσκονται στο μέσο όρο, είναι πολύ πιο ακριβά τα σπίτια των μεγάλων των μελών. Αυτό ισχύει για όλο το δημοτικό προσωπικό. Η αγορά έχει τις τιμές που έχει. Στο Χονγκ Κόνγκ 10 τετραγωνικά κοστίζουν όσο 200 τετραγωνικά σε κάποια μέρη της Ευρώπης. Παίρνουμε το μέσο όρο της αγοράς, το μέσο του πόσο είναι τα κρατημέλη, βγάζουμε ή προσθέτουμε ένα ποσοστό και έτσι προκύπτει το τι πληρώνουμε. Πάντοτε λαμβάνει υπόψη τι πληρώνουν τα κρατημέλη και παλεύουμε και είμαστε συνεχώς στο μέσο όρο. Φυσικά Πρόκειται περί πολλών χρημάτων. Κανείς αν το δει σαν νούμερο έτσι προκύπτει. Αλλά αν θέλει κανείς να έχει αντιπροσώπους παντού σε όλο τον κόσμο και κάπου που είναι ακριβή η στέγη, τότε κανείς θα πρέπει να πληρώσει πολλά. Θα τους δώσουμε τη διακριτική ευχέρεια, θα τους δώσουμε κάποιο καταβοκοπή ποσό, να αποφασίσουν τέλο πάντων οι υπαλλήλοι μα αν θέλουν να μείνουν σε μικρότερο σπίτι στο κέντρο ή να έχουν περισσότερο μεγαλύτερο σπίτι κάπου στα προάστια της πόλης που θα υπηρετήσουν και έτσι θα έχει περισσότερο περιθώριο το προσωπικό μας θα έχουν την επιλογή του που θα μείνουν και θα υπάρχει μια οροφή ανά βαθμό και αν, ανάλογα με τα καθήκοντα που ε, εκτελούν. Ε, απασχολούμε πολλούς τοπικούς της αντιπροσωπείας, τους αξιοποιούμε. 3.000 ε, τέτοιους υπαλλήλους τοπικούς έχουμε, δυνάμει του τοπικού κάθε φορά εργατικού δικαίου, σεβόμαστε τις συνήθειες απασχόλησης, ο δε μισθός τους βασίζεται στα όσα πληρώνει ο ΙΕ ανάλογα και άλλοι μείζονες οργανισμοί. Πώς θα το σύστημα να το αναθεωρήσουμε, να το κάνουμε κάπως περισσότερο ευέλικτο. Πάντως πρόσφατα ήρθαμε σε κάποια συνάντηση με αυτούς τους υπαλλήλους μας είπαν ότι έχει πέσει το δίκαιο τους επίπεδο εμείς ε, τους απαντήσαμε ότι αναζητούμε πάντα τους υποταλαντούχους, ότι είμαστε καλός εργοδότης και ενταγωνιζόμαστε τον ΟΗΕ και άλλα θεσμικά όργανα, οπότε αν θέλουμε να κρατήσουμε το ίδιο επίπεδο θα πρέπει να τους δώσουμε έναν λογικό μισθό. Όσον αφορά τώρα την επιλογή, επιλέγονται με δημοσιεύσεις, έχουμε διάφορο σύστημα ε, υποβολής επιτήσεων και επιλογής των υπαλλήλων και προσπαθούμε πάντοτε να επιλέξουμε τους άριστους. Δεν αναφέρεται τώρα για τα πάλι και τα οικονομικά του εσείς, κυρία Γκρέσλα και κάποιος άλλος. Να τα πάρουν τα από την αρχή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Αυτές που δεν μπορούν να ασκήσουν δεν μπόρεσαν στην αρχή τότε δεν μπορούσε να κάνει ο υπότος εκπρόσωπος ο κύριος Σολάνα Επίσης, σε κάποιες περιπτώσεις, πάρα πολύ χρήσιμο να έχει κανείς κάποιον ο οποίος να ασχολείται με ένα πρόβλημα περιφερειακό μόνο ή με ένα άλλο ζήτημα. Δεν μπορεί να το παρακολουθήσει δουλεύοντας μόνο γι' αυτό στην υπηρεσία. Έχουμε όμως τις ε, δασέ Ε, τον προπολογισμό που καλύπτει αυτά τα ζητήματα, οπότε και κατά αυτόν τον τρόπο έχουμε περισσότερη ευελιξία από ό,τι στον διοικητικό προπολογισμό και έτσι σε κάποιες ε, περιπτώσεις κρίσεων συγκροτούμε τέτοιες ε, ομάδες όταν δεν μπορεί ο σύνδεσης προπολογισμό να διαχειριστεί το να καλύψει αυτό το θέμα. Άρα υπάρχει συμπληρωματικότητα. Θα πρέπει όμως να υπάρχει και συνέργεια. Και αυτό προσπαθεί να πετύχει η ψήστη εκπρόσωπος, η πάτη εκπρόσωπος. Προσπαθούμε επομένω να δούμε πώς αυτά θα ενταχθούν στο προϋπολογισμό, όπως θα συνάδουν προς τον προϋπολογισμό που τα ξέρετε αυτά τα ζητήματα. Θα θέλαμε αυτό να είναι τμήμα, αυτά τα χρήματα που σας είπα είναι τμήμα του προϋπολογισμού μας. Ξέρω ότι αυτό προκαλεί ανησυχία, αυτό σημαίνει μια μεταφορά από το, από το τέταρτο στο πέμπτο κεφάλαιο και όσοι ξέρουν τις λεπτομέρειες του θέματος, αυτό είναι κάτι σαν μια αίρεση στο βασικό δόγμα. Έτσι καλώς και περί διοικητικού προπολογισμού. Αλλά όλα αυτά θα, ήταν, θα μπορούσαν να γίνουν. Ε, θα μπορούσε όμω κανεί αυτά όλα τα χρήματα τα έχει στον προπολογισμό μας, αλλά να μην αφήνει το περιθώριο να χρησιμοποιηθούν για κάτι άλλο. Άρα ο ειδικό εκπρόσωπο για αυτά τα ζητήματα μπορεί να έχει την ειδική προοικοδότηση. Και αυτό εξετάζουμε τώρα το πώ θα έχουμε την, την πιο αποτελεσματική λειτουργία. Το θέμα είναι περίπλοκο. Θα πρέπει αυτό να ξανασυζητηθεί. Τα δικρατημέλη Ξέρω ότι οι διπλωμάτες της υπηρεσίας μας συνεχίζουν να είναι υπόλογοι στην Πολιτική Επιτροπή. Αλλά από την άλλη μεριά θα πρέπει να, είναι, να υπάρχει κάποια ιεραρχία. Θα πρέπει να υπάρχει μια πολιτική ολοκλήρωση τέλο πάντων ιεραρχίας. Από την άλλη μεριά όμως έχουμε κάποια καθήκοντα, κάποιες κρίσεις όπου πρέπει να υπάρχει κάποιος που να ασχολείται με αυτές τις κρίσεις. Να, όπως έγινε με την Αραβική Άνοιξη. Σουδάν, Κεντρική Ασία, Κάφκασος, οπότε είχαμε κάποιες εκμένες προσωπικότητες που ασχολήθηκαν με αυτά τα προβλήματα. Ε, είναι καταρχήν ε, θέμα κλιματικότητας, αλλά είναι τα πράγματα περίπλοκα πλευράς δημιουργικής όσον αφορά τις συμβάσεις για την ασφάλεια, ασχολήθηκα δύο χρόνια με αυτό, και στην πρώτη έκθεση που υπέβαλα δεν είχα πιστεί ότι έχουμε την καλύτερη δυνατή διαχείριση. Όπως είπε η κυρία Γκρέσλη, είχαμε κάποιες υπερημερίες ε, όσον αφορά τι πληρωμές, κάποια προβλήματα με τις νέες συμβάσεις και προσπαθήσαμε πάρα πολύ και εμείς με τα προβλήματα. Δεν τα έχω όλα δει για φέτο. αλλά νομίζω θα άρω τι επιφυλάξει που είχα διατυπώσει για την περσινή χρήση και στη φετινή θα δώσω το πράσινο φω. Πέρσι το ελληνικό συνέδριο είχε επισημάνει κάποια προβλήματα. Είχαμε στη Βενεζουέλα ε, την ε, ανανέωση μια συμβάσεω επανειλημμένα χωρί διαγωνισμό. Οπότε θα πρέπει να δούμε το ότι αυτό γίνεται σε κάποιες αντιπροσωπείες, όχι λόγω κακής διαχείρισης, αλλά πολλές φορές είναι περίπλοκο σε κάποιες αγορές, κάποιες χώρες να γίνονται διαγωνισμοί. Οπότε λέει κανείς, αφού είναι τόσο δύσκολο, άντε ας ανανεώσουμε την ίδια σύμβαση, αφού δουλεύει καλά η υπηρεσία. Οπότε προσπαθούμε και εμείς να βάλουμε τάξη, να βοηθήσουμε τις αντιπροσωπείες και θα τα κάνουμε αυτά φέτος. Τώρα, για την Όλαφ, όπως ε, είπε και ο κύριος ε, Σαλαφράγκα, μόλις τελευταίες μέρες ε, λύσαμε τα τελευταία θέματα που εκκρεμούσαν με τον Τζοβάνι Κέσλα. Εντάξει, μπορεί να πήρε λίγες μέρες, πήρε κάποιες λίγες εβδομάδες. Και το θέμα ήταν κατά πόσο μπορεί η Όλαφ να διαβιβάσει κάποιους φακέλους στις δικαστικές αρχές τρίτων χωρών. Δεν θέλω να κατονομάσω τις χώρες, αλλά ας πούμε με κάποια χώρα όπου ακριβώς δεν κατησχεί το κράτος δικαίου. Θέλουμε διαφάνεια να ξέρουμε τι θα γίνει, να μην έχουμε στο έργο της Όλαφ, αλλά θέλουμε τα πράγματα να γίνουν σωστά. τέλο πάντων, τελικά τα βρήκαμε. Και τελικά στην πράξη 99% από αυτό το μνημόνιο κατανόηση, έκλεισε. Και από αυτού θα δουλεύουμε όπως και έχουμε δουλέψει τόσους μήνες. Οπότε το πήγαμε καλά τόσες υποθέσεις με την Όλαφ. Θα ζητήσω την Όλαφ να σας ενημερώσει κύριε Ντότσιν. Πάντως τα υπόλοιπα πρέπει να σας τα πει η ίδια η Όλαφ. Σε κάποιες περιπτώσεις έκλεισαν οι φάκελες, σε άλλες υπήρξε ανάληψη πειθαρχικών κυρώσεων ή επιβολή και σε κάποιες είχαμε συστώσεις και σε 12 έρευνε τέλος πάντων δεν συνέχεια και συνεργαζόμαστε σε στενά με την Όλαφ γίνεται καλή δουλειά. Και τώρα για το τελευταίο. Συγγνώμη που δεν το κατάλαβα πολύ καλά, αλλά νομίζω ότι είναι αυτό το οποίο λέμε αναστολή των λογαριασμών. Κύριε Πρόεδρε, και εγώ είχα το ίδιο ερώτημα επί του ιδίου ζητήματος. Ένας μηχανισμός του προϋπολογισμού που αφορά τη μεταφορά ενός κονδυλίου από τον ένα λογαριασμό στον άλλο. Ας πούμε, βγάζουμε κάτι από τις πληρωμές, μετά πληρώνουμε στις τοπικές αρχές το ΦΠΑ ή έχουμε κάποια γενικά επιδόματα για το προσωπικό, τα βγάζουμε, τα βάζουμε σε αυτό το, σε αυτό το αποθεματικό, ας το πούμε. Ε, είναι κάτι σαν ένας λογαριασμός που εκρεμεί μέχρι ότου συμβεί κάτι. Δηλαδή βοηθάει πάρα πολύ. Μπαίνουν χρήματα από εκεί και βγαίνουν όταν χρειάζεται. Είναι πάντως συνήθες πρακτική λογιστική. Το χρησιμοποιεί η Κομισιόν. ποια χρήματα που θα πρέπει κάπου να πάνε στην άκρη και να πληρωθούν κάπου αλλού κάποια στιγμή αργότερα. Ακούσαμε Επίσης τι είπε η κυρία Γκρέσλε για κάποιες υπερημερίες. Ε, αν κάνουμε κάποιο σφάλμα και αργήσαμε να καταβάλουμε κάτι, ε, τότε βεβαίως και έχουμε την υποχρέωση να καταβάλουμε κάποιους τόκους στον δικαιούχο. Όπως λέει η ερώτηση 29, Deutsche Telekom, Argos και κάποια άλλη εταιρεία, είναι περιπτώσεις περιπτώσεις κάποιων εταιριών παροχής περισσότερων ασφαλείας, αυτοί που προσέχουν τις πόρτες, δεν θα έπρεπε να είμαστε περίμενοι, αλλά συμβαίνουν αυτά. Δεν πληρώσαμε όταν έπρεπε, οπότε και ο αντισυμβαλόμενος δικαιούται τόκους υπερημερίας. Κάποιες αυτές οι εταιρείες είναι μεγάλες εταιρείες, κάποιες είναι λιγότερο μικρές αλλά για μικρομεσαίε επιχειρήσει που συναλλασσονται μαζί μα είναι σημαντική αυτή το υπέρημα. Τώρα, κύριε Αγγλισό, όσον αφορά του επικεφαλεί των αντιπροσωπιών και την γεωγραφική ισορροπία τη κατανομή, τι να σα πω. Δεν θεωρώ ότι τα στοιχεία ερμηνεύονται όπως τα είπατε εξή, αλλά συμφωνώ μαζί σας στο εξή. Πώς να σας το πω τα πιο πρόσφατα προσχωρήσαν τα κράτη-μέλη εκπροσωπούνται λιγότερο. Λέω για τους 10 που μπήκαν το 2004. Γιατί δεν έχουν ε, τόσο απόθεμα προσωπικού, το πούμε, όσο τα παλιότερα κράτη-μέλη που ξεκίνησαν την ιστορία του 1950. Αν κοιτάξει βαθμό υψηλόβαθμος υπαλλήλου, έχουμε 7 από τη Γαλλία, 6 από την Γερμανία, 3 από το Ηνωμένο Βασίλειο, που βρίσκονται στην τις ανώτατες θέσεις. Ερώτηση 16 ήταν αυτή. Τώρα επικεφαλής αντιπροσωπιών είναι προκειμένο από ό,τι φαίνεται. Η Γαλλία πρωταθλήτρια με 15, η Ιταλία με 14, η Γερμανία με 10, ακολουθεί κλπ. Με όλο το σεβασμό. Δεν ήταν θέμα πολιτικής επιλογής. Το θέμα ήταν τι ήταν πιο, πιο δόκιμο, πιο χρήσιμο υπάρχει αντικειμενικότητα και διαφάνεια σε αυτή τη διαδικασία. Όμω είναι αλήθεια και θυμάμαι πάρα πολύ καλά ότι το 2011 τότε που συγκροτηθήκαμε και που προσλάβαμε πάρα πολλού, είχαμε πολύ περισσότερες αιτήσει από Γάλλους διπλωμάτες από, από άλλη εθνικότητα. Ε, επιλέγουμε από τους υποβαλλόντες αιτήσει. Οπότε έτσι πάει. Κύριε Μίντερ. για τη συστέγαση αυτή που είπατε. Υπάρχει συνέργεια μεταξύ των μελών και της υπηρεσιοστηρής δράσης όσον αφορά τις προξενικές υπηρεσίες και το μελετούμε, εργαζόμαστε επ' αυτού και αυτό είναι περίπλοκο γιατί προσπαθούμε να συγχρονίσουμε την, την ατζέντα των κρατών μελών τις συμβάσεις μίσθος ακινήτων, τη... ό,τι συμβάσεις έχουν, τα υπηρεσίες εξωτερικών και... Α, πρόσφατα στην Αθήνα συνεργαστήκαμε με το ΙΠΕΞ είπαμε ότι θα πρέπει να δεσμευτούμε να συστεγαστούμε το κάτι το οποίο απαιτεί από εμάς να λάβουμε υπόψη τις ανάγκες των κρατών και τα κράτη-μέλη να πούνε ότι δεν θα μετακομίσουμε φέτος, να θα περιμένουμε φέτος να μετακομίσουμε τότε που εσείς θα ε, φρεσκάρτε το, το δικό σας κτίριο. και αυτοί θα βγουν κερδισμένοι, θα πάει η πρεσβεία τους σε καλύτερο κτίριο. Να πώς προκύπτουν οι δαπάνες με την πανωτική στρώα όσον αφορά τις προξενικές υπηρεσίες. Γίνεται αυτό. Να συνεργαστούν μαζί μας, στην υπηρεσία μας. Στο κτίριό μας τέλος πάντων. Στην Σαϊγκόνη, Χότζιμιν City, όπως τη λέμε σήμερα, εκεί Υπάρχει μια κοινή υπηρεσία που δίνει στη θεωρήση διαβατήριων για τις χώρες Σέγγεν από κοινού για όλες και αλλού. Έχουμε ξέρει στα κρατημένα ότι αν θέλουν μπορούν να μοιραστούν τη, τα γραφεία μας και να γίνει και εκεί το ίδιο όσον αφορά τις θεωρήσεις διαβατηρίων. Αυτό το πνεύμα διαπνέει το τι κάνουμε για να προβάλλουμε ένα κοινό πρόσωπο, κοινή βιτρίνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το γραφείο της αντιπροσωπείας μπορεί να το χρησιμοποιήσουν οι διπλωμάτες ε, ε, άλλων χωρών, τρίτων, που με επισκεφθεί αυτή τη χώρα. Ε, οπότε βλέπετε ότι εκεί πέρα κάνουμε πολλά. Τώρα, τι άλλο είπε ο κ. Σαραφράγκα. νομίζω απάντησε για την Όλαφ. Και το θέμα τώρα WLAD το λένε οι συνάδελφοι της ΔΕΦΚΟ. Πώς καλύπτονται από τον προπολισμό τα έξοδα των αντιπροσωπιών. Έχουμε τώρα τον κύριο Ντεμέλο, νέος Γενικός Διευθυντής. Θα πρέπει να προσαρμόσουν τον προγραμματισμό πριν την ολοκλήρωση του MFF με τη σημερινή κατάσταση. Δεν είναι τόσο μεγάλη η διαφορά στην κατάσταση, αλλά θα πρέπει να κάνουμε κάποιες προσαρμογές. Ας πούμε έχουμε το εργαλείο εταιρικής σχέσης. Χρειαστήκαν παραπάνω προσωπικό, αλλά θα πρέπει να δούμε, δεν μπορεί να διορίζουν παλιούς τη μια εβδομάδα για να τους απολύουμε την επόμενη. Για τον Παναμά να έχει ληφθεί υπόψη αυτό το οποίο είπατε, είναι περίπλοκο και αυτό το να ανοίγουμε και κλείνουμε την προσωπία, αλλά νομίζω ότι έχουμε λάβει το μήνυμα, ξέρουμε θέλει το κοινοβούλιο και ξέρουμε πώς θα ανταποκριθούμε. Τέλος δε, όσον αφορά τα θέματα τη παρακολούθηση και τη ασφάλεια. ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά τα παραπάνω εκατομμύρια που το κοινοβούλιο ενέκρινε να πάρουμε για φέτο και πάρα πολύ σοβαρά κοιτάμε πώς θα τα αξιοποιήσουμε καλύτερα και η βασική μας δε προτεραιότητα είναι στην επιλογή των ε, αντιπροσωπιών τόσο ώστε να μπορούμε να έχουμε ασφάλεια στις συνομιλίες και να έχουμε συνεδριάσεις που δεν θα παρακολουθούνται. Και όσον αφορά την κινητή τηλεφωνία και τη σταθερή τηλεφωνία, καλά δεν λέω, δεν, δεν έχω ψευδεστήσεις ότι όλα αυτά μπορούν να, να, να, να, να είναι αδιαπέραστα από την τεράστια πρόοδο της τεχνολογίας όχι μόνο των φίλων Αμερικανών αλλά και άλλων που έχουν λιγότερο άγαθες προθέσεις. Πρόκειται για ένα τομέα στον οποίο θα πρέπει να επιφέρουμε πολύ σημαντικές βελτιώσεις. Οπότε σας ευχαριστώ πάρα πολύ που εσείς ήσασταν πρωτοπόροι στο να βοηθήσετε με τα επιπλέον χρήματα και έτσι να κάνουμε κάτι ήδη από φέτος. Προσπάθησα, ε, Πρόεδρε, να απαντήσω σε όλα. Αν κάτι ξέχασα, ευχαρίστω να συμπληρώσω. Ευχαριστώ κύριο Σάλιβαν, λέει ο πρόεδρος Τόιρερ. Είναι σχεδόν αδύνατο βέβαια να ικανοποιήσει κανείς όλα τα μέλη της ε, κοινοβουλευτική Επιτροπής. Αλλά αυτό κάπου εντάσσεται και στην φύση των θεμάτων με τα οποία ασχολούμεθα. Η κυρία Κρέσλε, ωστόσο, έχει μια συμπληρωματική ερώτηση. Όχι, μην το λες αυτό. Αν θέλει κανείς, μπορεί. Ασχολούμεθα ιδιαίτερα με αυτό το νέο παιδί, διότι δεν γνωρίζουμε αρκετά γι' αυτό. Και γι' αυτό νομίζω ότι είναι και καλή η είδηση ότι όχι μόνο ασχολούμαστε όλοι με αυτό, αλλά και ότι έχουμε, διαβάσει τις σχετικές εκθέσεις. Επανέρχομαι λοιπόν στο θέμα του top management. Λέτε ότι δεν έχετε τα σχετικά νούμερα. Ούτε εγώ τα έχω. Και γι' αυτό κάθισα και μέτρησα μόνη μου. Και κοιτάξτε, οι άνω πάνω πάνω θέσεις είναι όπως σας τις είπα. Αν έχετε άλλα νούμερα να μας τα δώσετε γιατί τα νούμερα που είπατε μετά από τις ερωτήσεις μας είναι σε πολύ ευρύτερη βάση γιατί αναφέρονται σε ολόκληρη την ε, υπηρεσία. Ωστόσο έχω δύο παρακλήσεις. Κάνετε και μία ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων ως Chief Operating Officer. Officer. Ξαναρωτώ γιατί άραγε καταργείται η θέση σας ή ποιος θα κάνει, ποιος θα ασκεί τα δικά σας καθήκοντα. έχουμε και τις σχετικές συμβάσεις μίσθωσης των κτηριών σας ή κατοικιών. Για μένα αυτό, η δική μου λίστα δηλαδή που έχω είναι μεγάλη. Στην προ προηγούμενη έκθεση είχαμε και, θα, θα πρέπει να δούμε και τις ε, ε, οικονομικές εκθέσεις, τις εκθέσεις οικονομικού ελέγχου. Τώρα, για τα θέματα του προσωπικού. Κάνετε μια staff review, την οποία δεν λαμβάνουμε. Θεωρώ έντιμο εκ μέρους σας να μας υποβάλλετε και αυτά τα νούμερα, εφόσον τα έχετε. Υπάρχει staff report της υπηρεσίας, την οποία δεν λαμβάνουμε εμείς. Θα ήθελα λοιπόν να αντιλάβουμε. λάβουμε. Πρόεδρος Τόιρερ, ευχαριστώ. Να απαντήσετε παρακαλώ για το πρώτο σας θέμα. Έλεγα ότι εξαρτάται πώς μετράτε τα νούμερα του senior management. Εγώ μιλούσα για διευθυντές και άνω. Αν τώρα στενέψετε πιο πολύ την πυραμίδα, κοιτάξτε, Κάπω πάντα θα υπάρχει, διακόπτη κυρία δεν την ακούμε, πάντα θα υπάρχει κάποια έλλειψη ισορροπία. Αλλά και αυτό βεβαίως κυμαίνεται, άλλοι φεύγουν, άλλοι έρχονται. Υπάρχει κίνηση, ε, οι συμβάσει πρόκειται να ανανεωθούν το πρώτο τρίμηνο του επομένου έτους, άλλοι προ, ε, προάγονται και ο διάδοχος της κάθε άστον ίσως θα θέλει κάνει κάποιες αλλαγές. Δεν είναι στατική η κατάσταση. η κατάσταση από άποψη στατική πάντα θα έχει κάποια έλλειψη ισορροπίας. Αν ε, ε, λάβετε ένα ενσταντανέ οποιαδήποτε στιγμή θα βρείτε κάποια έλλειψη ισορροπίας και αν ξανακάνετε την ίδια καταγραφή μετά από δύο χρόνια θα δείτε πάλι κάποιες αλλαγές. Άρα χρειάζεται κάποια προσεκτικότερη εξέταση μέσα σε ένα βάθος χρόνου. Υπάρχει μια ποικιλότητα. Σε ό,τι αφορά το πόσο απαραίτητος δίθεν είμαι κυρία Κρέσλε, νομίζω ήταν σημαντικό στα αρχικά στάδια ο Πιέρ και εγώ να κάνουμε μια κατανομή έργου που νομίζω ότι πράγματι ορισμένοι δεν συμφώνησαν με τον τρόπο που το κάναμε αλλά θα ήταν πολύ δύσκολο ή οσδήποτε εξημών ή τέλο πάντων ή ο ένας ή ο άλλος να κάνουμε ολόκληρη τη δουλειά δηλαδή να είμαστε Executive Secretary General, δηλαδή να έχουμε τι επαφέ με το ε, Συμβούλιο ε, Υπουργών Εξωτερικών, ταυτόχρονα ε, τις επαφές με το Κοινοβούλιο και να διοικούμε όλο το σύστημα. Γι' αυτό χρειαστήκαμε ένα είδος δικέφαλης ε, ηγεσίας. Τώρα που το σύστημα έχει ξεκινήσει και προχωρεί και αν θέλει κανείς να εξορθολογήσει όπως είπε η Κάθη αλλά και πολλοί από εσάς άλλωστε λίγο σαν μεξικάνικο στρατός ε, δηλαδή πολλοί στρατηγοί και λίγοι στρατιώτες είναι βεβαίως και μια δυνατότητα να συγχωνευτούν οι δύο θέσεις σε μία θα χρειαστεί βεβαίως κάποια αναδιάρθρωση κάποια αναδιάταξη των μηχανισμών. Θα βρεθεί τρόπος να γίνει αυτό. Ε, για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, άμα καθίσω μια ώρα μπορώ να το φτιάξω το σχέδιο αυτό. Αλλά θα το εγκρίνει βέβαια ο διάδοχος της κάθε Άστον, γιατί η appointing authority είναι εκείνη που εγκρίνει ε, και αποφασίζει ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να γίνει η αναδιάταξη αυτή των ροών των υπευθύνων και επίσης ε, της κίνησης από την ύπατη εκπρόσωπο προς ε, τα κατώτερα επίπεδα του προσωπικού της. Με συγχωρείς ε, να δω μια στιγμή εδώ. Α, για, για τις τοποθεσίες, για τη location. Δεν τα λέει νομίζω αυτά δημοσιονομικός κανονισμός, νομίζω εγώ μου λένε όμως ότι μπορούμε να ε, περιλάβουμε μια στήλη ακόμη που να περιλάβει τα δεδομένα αυτά τα οποία ζητήσετε εάν θεωρήσει το Κοινοβούλιο ότι του είναι αναγκαία. Όπως ανεγνώρισε ο κ. Σαλαφράνκα δεν έχουμε τίποτε να κρύψουμε, μπορούμε να ανοίξουμε όλα μας τα βιβλία. Ο μόνος περιορισμός είναι οι δυνατότητες του προσωπικού να κάνουν τη δουλειά αυτή. Οι πόροι που διαθέτουμε. Μα το κάνετε ούτως ή άλλως. Δίνετε τις προφορίες αυτές. Στην πρώτη έκθεση το κάνατε, στη δεύτερη έκθεση τα δώσατε. Μόνο, ναι, προσπαθούμε να βασιστούμε σε βέλτιστες πρακτικές. Δεν είναι καν πρόσθετος, πρόσθετος φόρτος εργασίας. Και μπορείτε να προσθέσετε ότι πρόκειται η οικειοθελή υποβολή ε, δεδομένων, λέει ο πρόεδρος Τόιρερ. Σα ευχαριστώ λοιπόν, ωραία, για να ολοκληρώσουμε τώρα την συζήτηση. Κοιτώντα λίγο και το ρολόι, να δώσω το λόγο πάλι στο ελεγκτικό συνέδριο, εφόσον το επιθυμούν, και μετά στον εισηγητή. Ο κύριος Μουγκουρούζα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συνοπτικά μπορεί να πει κανείς ότι τα μόνα ευρήματά μας σε σχέση με την υπηρεσία εξωτερικών δράσεων φέτος αναφέρονται στην ενημέρωση των καταστάσεων προσωπικών και οικογενειακών του προσωπικού για την καταβολή των επιδομάτων. Δεύτερον, για τα πιο σοβαρά ευρήματα που είχαμε πέρσι, γνωρίζουμε ότι η υπηρεσία ήδη βρίσκεται στη διαδικασία αντιμετώπισης τους και θα είμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε τις αλλαγές αυτές όταν θα προβούμε στο μέλλον στους οικονομικούς ελέγχους, όπως είπα σε εναλλακτική βάση των συστημάτων εποπτείας και ελέγχου της υπηρεσίας. Και κάνουμε βέβαια και την εξέταση του follow-up που δίνεται στις συστάσεις μας. Θα ήθελα επίσης να κάνω ένα σχόλιο για δική σας ενημέρωση σχετικά με τις συντάξεις. Είναι σαφές και λέχθηκε ήδη δεν είναι ειδικό χαρακτηριστικό της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης. Σας, βιβλιορώ, σας πληροφορώ λοιπόν ότι στα πλαίσια των δηλώσεων αξιοπιστίας 2014 το ελεγκτικό συνέδριο αξιολογεί τους τρέχοντες υπολογισμούς για τις συντάξεις για να περιληφθεί στον ισολογισμό της Ένωσης το επεξεργαζόμαστε λοιπόν αυτό. Και τέλος, όπως είπε ο συνάδελφός μου Φαζάκας, το συνέδριο θα μπορέσει να προσθέσει και άλλες πληροφορίες για την αποδοτικότητα της υπηρεσίας όταν θα έχουμε συντάξει την ειδική μας έκθεση. Τίποτε άλλο. Ευχαριστώ. Και τώρα εσείς κύριε Ταμάς Ντόιτς ως εισηγητής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμη κύριε Διευθυντά και εσείς κύριε και κύριοι συνάδελφοι είμαι σύντομος. Νομίζω ότι ήταν χρήσιμη η συζήτηση. Ήδη είπα από την αρχή της ότι επιθυμώ να ευχαριστήσω τον κύριο Σάλιβαν καθώς και τους συνεργάτες του για το ότι μπορέσαμε να λάβουμε λεπτομερείς απαντήσεις στις ερωτήσεις μας. Δεν είναι απλά μια έκφραση αυροφροσύνης. Θεωρώ ότι εμείς οι βουλευτές έχουμε σημαντική ευθύνη. Θέσαμε λοιπόν με ευθύνη τις ερωτήσεις μας και λάβαμε απαντήσεις. Και ο στόχος μας είναι να βελτιωθεί η ποιότητα της εκθέσεως. Ευχαριστώ. Ο πρόεδρος Τόιρερ. Ευχαριστώ και εγώ σας κύριε Σιγητά. Και εδώ ολοκληρώνεται η συζήτηση του θέματος αυτού και ευχαριστώ και εσάς κύριε ο Σούλιβαν και σας ευχαριστώ, όπως, σας ευχαριστώ και σας παρακαλώ να διαβιβάσετε τους χαιρετισμού μας στην ε, ύπατη εκπρόσωπο την οποία ελπίζουμε να δούμε σε ένα επόμενο στάδιο ή δεμή των ή την ε, διαδοχό της. Ο πρόεδρος Τόιρερ, ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και με την άδειά σας να προχωρήσω στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Πρόκειται για την έκθεση Μπαλσίτης για την ειδική έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου για τους εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας παρακαλώ βεβαίως να αποχωρήσετε όσοι το επιθυμείτε με ησυχία και σε τρόπον ώστε να μπορέσει να μιλήσει ο εισηγητής Μπαλσίτης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν είναι η πρώτη φορά που ασχολούμεθα με το ζήτημα αυτό στην Επιτροπή μας. Ο Ντέρ Βόγκαν είχε προτιμάσει στο παρελθόν ένα έγγραφο εργασίας που είχε να κάνει με την ειδική αυτή έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου όσον αφορά τους εργαζόμενους με καλύτερης ηλικία. Το έγγραφο αυτό θα θυμάστε ότι είχε εντοπίσει τότε ένα συγκεκριμένο αριθμό προβλημάτων τα οποία ουσιαστικά παντλαμβάνονται, υφίστανται, εξακολουθούν και υφίστανται και εντοπίζονται και στο δικό μου το έγγραφο. Πώς δηλαδή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το ESF, προκειμένου να καταφέρουμε να ευνοήσουμε λίγο περισσότερο και να στηρίξουμε τους ηλικιωμένους εργαζομένους. Ξέρετε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο έχει ως στόχο να υποστηρίξει κυρίως τους ανέργους, καθώς επίσης ε, και τις μειονεκτούσες ομάδες ε, του πληθυσμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι δαπάνε που γίνονται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στην τελευταία περίοδο προγραμματισμού 2007-2013 ανέρχονται σε 75 δισεκατομμύρια ευρώ, 17% δηλαδή του συνόλου του προϋπολογισμού. Όταν λοιπόν αναφερόμαστε στα προβλήματα αυτά τα οποία έχουν προκύψει με την εφαρμογή των επιμέρους προγραμμάτων, βλέπουμε καταρχάς ότι ε, δεν υπάρχει συνεκτικότητα και δεν υπάρχουν αξιόπιστα δεδομένα από τα κράτη-μέλη. Στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να μας δώσουν συγκεκριμένα στατιστικά δεδομένα για το πώς οι τελικά ηλικιωμένοι εργαζόμενοι κατάφεραν να αποκτήσουν νέα, νέες επαγγελματικές γνώσεις ή αν κατάφεραν τελικά να έχουν πρόσβαση σε μια νέα θέση εργασίας. Θα ήταν πολύ θετικό να είχαμε τους απαραίτητους δείκτες οι οποίοι θα μας επέτρεπαν πραγματικά να δούμε πόσο αποτελεσματικό είναι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για τους εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας και αν τελικά οι κοινοτικοί πόροι δαπανώνται σωστά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την πλευρά της είναι υπεύθυνη για την χρηματοδότηση αυτή, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και για τον κοινοτικό βέβαια προπολογισμό. και είναι αυτή η οποία θα πρέπει να καταρτήσει ένα σύστημα συλλογής αξιόπιστων δεδομένων από τα κράτη-μέλη. Αν λάβουμε τώρα υπόψη μας τις συστάσεις που κάνει το ελεγκτικό συνέδριο στην έκθεσή του και που έχω συμπεριλάβει και εγώ στο σχέδιο ψηφίσματος, βλέπουμε ότι πρώτον θα πρέπει να καταρτιστούν ειδικοί δείκτες στα προγράμματα, τα λειτουργικά προγράμματα, θα πρέπει να υπάρχει σχέση αιτίου και αιτιατού ανάμεσα στις χρηματοδοτούμενες δράσεις και τους στόχους που θέλουμε να πετύχουμε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να γίνει λίγο πιο αποτελεσματική στην ε, διασφάλιση της παρακολούθησης των προγραμμάτων, προκειμένου αυτά εν ευθέτω χρόνο να διορθωθούν. Αν δούμε δηλαδή κάποια στιγμή ότι δεν επιτυγχάνουμε τους ευκταίους στόχους μέσω των προγραμμάτων αυτών. Ακούσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι ε, γνωρίζουν ότι ήδη υπάρχουν κάποια προβλήματα, ότι έχουν καταφέρει πολλά από τα προβλήματα αυτά να τα διορθώσουν για τη νέα περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, ωστόσο όμως υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες για το αν θα καταφέρουμε τελικά να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά στην επόμενη περίοδο προγραμματισμού. Πολύ φοβούμαστε δηλαδή ότι θα καταλήξουμε πάλι σε ένα πολύπλοκο σύστημα με πάρα πολλά διαφορετικά έγγραφα, τα οποία δεν θα μας προσδίδουν τα απαραίτητα αξιόπιστα δεδομένα, τα οποία θα μας επέτρεπαν να λάβουμε κάποιες σωστές αποφάσεις όσον αφορά τα προγράμματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Καλό λοιπόν για άλλη μια φορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταρτήσει τις βασικές αρχές για τη συλλογή των δεδομένων και ένα σύστημα συλλογής δεδομένων. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε συνάδελφε. Μπορεί να αρχίσει η συζήτηση τώρα η κυρία Ορτής Βιλέγια. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα ήταν το δημογραφικό για τις βιομηχανικά ε, προχωρημένες χώρες. Οπότε υπάρχει έθιμα στο εξωτερικό και οπότε θα πρέπει για την πολιτική απασχόληση να δούμε τι γίνεται όσον αφορά του εργαζομένου πάνω από τα 55 και σε εθνικό και σε γενικό επίπεδο. Και ένα από του στόχου ήταν να μπορέσουμε να δούμε πώ θα αντιστρέψουμε την, την ροή των πραγμάτων. Ε, Βεβαίω, Φυσικά και μπορεί οι άνω των 55 εργαζόμενοι να δώσουν προ την αξία σε επιχειρήσει. Έχουμε επομένω την πρόσφατη κρίση τη απασχόληση και άρα θα πρέπει να δούμε ότι πώ μπορούν να βοηθήσουν όσον αφορά την αύξηση τη ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων ε, με τις γνώσεις και την εμπειρία τους. Επίσης θα πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι ο στόχος της στρατηγικής για το 2020 είναι ο ρυθμός της απασχόλησης να ανέβει πάνω από το 75% και γι' αυτό πρέπει αυτοί οι εργαζόμενοι να ενταχθούν στην αγορά εργασίας το οποίο θα είναι πάρα πολύ σημαντικό και επ' αυτού έχει εργαστεί ε, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Να μην ξεχνούμε όμω ότι δεν είναι γραφείο εργασία το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Φτιάχνει κάποια προγράμματα ούτω ώστε να δίνει περισσότερε προοπτικέ για χιλιάδε εργαζομένου. Οπότε το πρόβλημα κατά τη γνώμη είναι να δούμε πώ θα επισημανθούν οι σωστοί δείκτε ούτω ώστε να μπορέσουμε να δούμε πώ αυτά τα μέτρα θα είναι πιο αποτελεσματικά και πώ θα κατευθύνονται καλύτερα οι σχετικέ δαπάνε. Ε, του, Ταμείου. Και οπότε έχει αρμοδιότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπληρωματική της αρμοδιότητας των κρατών μελών. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να μένουν αδρανείς σε σχετικές διατάξεις και γι' αυτό θα πρέπει να επισημάνουμε τους κοινούς δείκτες, να τους εφαρμόσουμε και έτσι να ληφθούν τα, τα μέτρα πρέπει και οπότε θα πρέπει να δούμε ότι η πολιτική επασχόληση καλύπτει το σύνολο των κρατικών δράσεων προς την κάλυψη του ε, ε, ενεργού πληθυσμού για λογαριασμό άλλου. Και οπότε έτσι θα πρέπει να δούμε πώς θα παραταθεί ε, η ενεργή περίοδος της ζωής αυτών των προσώπων και θα πρέπει να δούμε πώς θα έχουμε κοινωνικές συνθήκες που θα είναι ευμενείς προς τούτο και θα έχουμε, να έχουμε τελικά αποτελέσματα από τα 2013 κάποιο που να πετύχαμε. Έχουμε το νέο κώδικα διοντολογία στην Ευρώπη για την αρχή του συνεταιρίζεστε. Το αυτό απαιτεί από τα κράτη-μέλη να ενισχύσουν τη συνεργασία του και να συνεργαστούν οι αρμόδιες αρχές όσον αφορά τους πόρους του διαδικών ταμείων και βεβαίως θα πρέπει οι πληροφορίες, οι καλές πρακτικές, όλα αυτά να τα μοιάζουν τα κράτη-μέλη και έτσι να κάνουν αποτελεσματική χρήση των ε, ταμείων σε την περίοδο του προγραμματισμού για την περίοδο 2014-2020. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Από τις άλλες πολιτικές ομάδες επιθυμεί κάποιο μέλος να λάβει θέση, όχι, από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο κ. Κέρσμακερ. Ελπίζω σωστά να προφέρα το όνομά σας. Πολύ καλά κύριε Πρόεδρε, πολύ καλά. Και σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Να ευχαριστήσω τον εισηγητή για αυτό το σχέδιο έκθεσης, το οποίο πραγματικά περιλαμβάνει κάποιες πολύ σημαντικές συστάσεις, προκειμένου να καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε καλύτερα το ζήτημα των ηλικιωμένων εργαζομένων και της παράτασης του επαγγελματικού βίου. Πρέπει να σας πω ότι είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες για τη δουλειά που έχει γίνει από το λεκτικό συνέδριο, γιατί πραγματικά έχει καταφέρει να εντοπίσει κάποιες αδυναμίες, τι οποίε πρέπει να βελτιώσουμε για να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα των ηλικιωμένων εργαζομένων. Τώρα, ποια είναι τα συμπεράσματα τη έκθεση του λεκτικού συνεδρίου. Ουσιαστικά η έκθεση αυτή αναφέρεται στο εφιστάμενο ρυθμιστικό πλαίσιο. Το πλαίσιο αυτό δηλαδή που είχε να κάνει κυρίω με την περίοδο 2007-2013. Όντω, ο παλαιότερος αυτός κανονισμός, γιατί ξέρετε ότι από την 1η Ιανουαρίου έχει αρχίσει να ισχύει ένας νέος κανονισμός για τη νέα περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, ο παλαιότερος λοιπόν αυτός κανονισμός δεν προέβλεπε έναν ορισμό για τον εργαζόμενο μεγαλύτερης ηλικίας, για τον ηλικιωμένο εργαζόμενο. Ποιοι ήταν οι άνθρωποι αυτοί. Κάθε κράτος μέλος είχε το δικό του ορισμό. Επίσης δεν υπήρχαν κοινοί δείκτες στα πλαίσια του προηγούμενου ρυθμιστικού πλαισίου, πράγμα το οποίο επιδίδωνε πάρα πολύ, επιδίδωνε πάρα πολύ το έργο της παρακολούθησης, αν θέλετε, της σχετικής πολιτικής. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι στα πλαίσια του προηγούμενου κανονισμού όλοι οι εργαζόμενοι ουσιαστικά μπαίνανε σε πάρα πολύ γενικές κατηγορίες, πολιτικές δηλαδή γενικές για την απασχόληση ή συγκεκριμένα μέτρα τα οποία μπορούσαν να είχαν να κάνουν μόνο με κάποια τμήματα του πληθυσμού, εν προκειμένου τους ηλικιωμένους εργαζομένους. Αυτή τη στιγμή έχουμε πολιτικές που απευθύνονται πλέον σε όλους τους εργαζομένους, αλλά δεν υπάρχουν όντως συγκεκριμένε πολιτικές για τους πιο ηλικιωμένους εργαζομένους. Τώρα, στην έκθεση του εκτικού συνεδρίου γίνονται συγκεκριμένε συστάσεις, οι οποίες έχουν ληφθεί υπόψη στο νέο ρυθμιστικό πλαίσιο, και καλύπτεται όντως η περίοδος προγραμματισμού 2014-2020. Η πρώτη σημαντική αλλαγή που έχει επέλθει με τον νέο αυτοκανονισμό... είναι το ότι οι πόροι πλέον που διαθέτουμε και στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου θα εστιάσουν περισσότερο στην στρατηγική Ευρώπη 2020 και τους βασικούς στόχους που αυτή εμπεριέχει κυρίως για την απασχόληση, ιδίως αν θέλουμε να αυξήσουμε την απασχολησιμότητα σε επίπεδο 75%, προφανώς πρέπει να στοχεύσουμε και στους ηλικιωμένους εργαζομένους. Γι' αυτό το λόγο στο νέο κανονισμό θα δείτε ότι μία από τις σημαντικές προτεραιότητες χρηματοδότησης έχει ως στόχο κυρίως τους μεγαλύτερους εργαζομένους, εργαζομένους μεγαλύτερης ηλικίας. Μια άλλη σημαντική καινοτομία του νέου κανονισμού όπου βασιζόμαστε βασικά εδώ και στην εμπειρία που έχουμε από το προηγούμενο κανονισμό, είναι ότι οι επιδόσεις πλέον θα ελέγχονται και θα αξιολογούνται με πιο σφαιρικό τρόπο. Θα έχουμε στο πυρήνα, στην καρδιά του νέου προγράμματος, ένα πραγματικό σύστημα αξιολόγηση των επιδόσεων. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να λένε ακριβώς τι έχουν επιτύχει, ποιους στόχους έχουν, επιτύχει, με ποιο τρόπο και πότε. Και αυτό μας οδηγεί σε μια άλλη σημαντική καινοτομία το ότι θα αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε πλέον κοινού δείκτες όσον αφορά τα αποτελέσματα. Δείκτες οι οποίοι θα χρησιμοποιούνται για όλα τα προγράμματα και θα μας βοηθήσουν να παρακολουθούμε καλύτερα τις επιδόσεις των κρατών μελών. Αν πραγματικά δηλαδή τα προγράμματα λειτουργούν όπως θα έπρεπε να λειτουργούν. Οι δείκτες αυτοί έχουν καταρτιστεί μετά από μια ενδελεχή ανάλυση που έγινε με τη συνεργασία πολλών κρατών μελών κατά τη διάρκεια δύο ετών και καταφέραμε να καταλήξουμε σε αυτούς τους κοινού δείκτες ε, αποτελεσμάτων. Και οι δείκτες αυτοί αναφέρονται και στους ηλικιωμένους εργαζόμενους. Μία άλλη σύσταση, τέταρτη κατά σειρά στην έκθεση του Εκτικού Συνεδρίου, ζητά από τα κράτη-μέλη να θεσπίσουν τους απαραίτητους μηχανισμούς προκειμένου να έχουν ένα καλό σύστημα παρακολούθησης εποπτείας των προγραμμάτων και θα πρέπει να υπάρχουν και απαραίτητοι πόροι γι' αυτό. Και τέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει συνεχείς επενδύσεις προκειμένου να υπάρχει καλύτερη δυνατή καθοδήγηση του προσωπικού της αλλά και των συνεργαζόμενων που έχουμε στα κράτη-μέλη προκειμένου να έχουμε καθοδηγητικά αν θέλετε έγγραφα τα οποία θα χρησιμοποιούνται στα προγράμματα αυτά και εδώ περιλαμβάνεται και η διοργάνωση σεμιναρίων για τους συναδέλφους μας καθώς επίσης και τους συνεργαζόμενους από τα κράτη-μέλη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Επιθυμεί το ελεγκτικό συνέδριο να προσθέσει κάτι από ό,τι φαίνεται όχι. Αν λοιπόν τώρα ο εισηγητής ενδεχομένως επιθυμεί να προβεί σε τελικά σχόλια. Ναι, σύντομα κύριε Πρόεδρε. Επιθυμώ να ευχαριστήσω το ελεγκτικό συνέδριο για τις ε, ορθές συστάσεις, καθώς επίσης την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μας ικανοποίησε λέγοντας ότι θα υιοθετήσουν διαφορετικό σύστημα με δεσμευτικούς δείκτες έτσι ώστε να αποφευθούν παρόμοια προβλήματα στο μέλλον γιατί είναι περίεργο που από το 2007 έως 2013 δαπανήθηκαν αρκετά σημαντικά ποσά και εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε τα ίδια προβλήματα. Δεν έχουμε υποχρεωτικούς δείκτες, δεν είχαμε μέχρι τώρα. Δεν είχαμε απλό μηχανισμό μέτρησης για να, πούμε, να δούμε ποιες, ποια είναι η αποτελεσματικότητα των ταμείων. Από το 2014 και μετά θα πρέπει να ζητούμε να υπάρχει αυστηρή λογοδοσία για την διαχείριση των ταμείων σε όλες τις χώρες μέλη εφόσον πρόκειται για χρήματα των Ευρωπαίων πολιτών, των φορολογουμένων. Ευχαριστώ λοιπόν. Ευχαριστώ λέει και ο πρόεδρος Τόερελ Άρα και αυτό το θέμα εδώ λύγει. Θα προτείνω ένα σύντομο πεντάλεπτο διάλειμμα για να αναπαυθούμε και λίγο και αναμένουμε το Γενικό Γραμματέα και τον Αντιπρόεδρο στις 5 ακριβώς. Ε, σε λίγα λεπτά.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

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, επαναλαμβάνουμε την συνεδρίαση που διακόπη για λίγα λεπτά και απευθύνω το καλώς ορίσατε στον Γενικό Γραμματέα του Κοινοβουλίου κύριο Βέλε. Καλώς ήρθατε. Ο Αντιπρόεδρος Πιτέλα δυστυχώς έχασε την πτήση του, όπως μόλις άκουσα δεν θα μπορεί λοιπόν να παραστεί σήμερα. Άρα κύριε Βέλε θα πυροδοτήσουμε ακόμα εντατικότερα πυρά καθημών. Ας αρχίσουμε λοιπόν πρώτα ακούγοντας το ελεγκτικό συνέδριο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το 2012 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μαζί με το Συμβούλιο ελέγχθηκε από το ελεγκτικό συνέδριο. Εν προκειμένου θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι το ελεγκτικό συνέδριο δεν βρήκε σημαντικές ελλείψεις στο σύστημα εποπτείας και ελέγχου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ούτε έγιναν παρατηρήσεις για την πρόσληψη ε, συμβασιούχων ή άλλων υπαλλήλων του ε, Κοινοβουλίου. Ορισμένες ελλείψεις όμως βρέθηκαν στα συστήματα προμηθειών, τα οποία οφείλονται κυρίως σε διοικητικά σφάλματα, σε μια περίπτωση στην διαχείριση της διαδικασίας προμήθειας και σε άλλη περίπτωση κατά εφαρμογή άλλου κριτηρίου. Επίσης η καταβολή κοινωνικών επιδομάτων σε μέλη του προσωπικού, όπου σε παλαιότερα χρόνια είχε κάνει σχετικές παρατηρήσεις το ελεγκτικό συνέδριο, για το 2012 διεπίστωσε ότι το Κοινοβούλιο εφήρμοσε μέτρα για να μετριάσει το ενδεχόμενο αυτό. Ωστόσο, ο κίνδυνος να καταβληθούν αδικαιολόγητα επιδόματα παραμένει, διότι το σύστημα βασίζεται σε δηλώσεις των ίδιων των μελών του προσωπικού. Οι παρατηρήσεις για το 2012 περιλαμβάνουν επίσης ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να βελτιώσει τις διαδικασίες προμηθειών με κατάλληλους ελέγχους και καλύτερη κατεύθυνση, guidance. Γνωρίζει το συνέδριο ότι έχει αναλυθεί δράση και εκπαιδευτικά σεμινάρια και χορήγηση συμβουλών στις ε, εμπλεκόμενες υπηρεσίες και το συνέδριο θα παρακολουθήσει τη σχετική πρόοδο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και είμαι στη διάθεσή σας για η αντίποτε απάντηση ή διευκρίνηση ενδέχεται να επιθυμείτε. Πρόεδρος Τόιρερ, ευχαριστώ κύριε Μπογκουμούζα. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Βέλε. Ο Γενικός Γραμματέας. Πρώτα, για το 2012 γενική παρατήρηση και έτσι και για το πλαίσιο που καθορίζει το έτος αυτό. Από το 2012 βρισκόμαστε σε ιδιαίτερη κατάσταση σχετικά με τον προϋπολογισμό. Τα έτη 2012 και 2013 έχουμε αύξηση των ιδίων πόρων μας της τάξης του 1,9% και για το 2014 0,4%. Αυτό σημαίνει ότι τα κονδύλια μας σε πραγματικές αξίες μειώνονται από το έτος 2012. Αυτό ισχύει ιδιαίτερος εάν σκεφτεί κανείς ότι προσθέθηκε και το 28ο μέλος, η Κροατία, και ότι βεβαίως υπάρχουν ειδικέ δαπάνες που συνδέονται με το τέλος της κοινοβουλευτικής θητείας και με την προπαρασκευή της ε, εκστρατείας ενημέρωσης της κοινή γνώμης. Εκτός αυτού, όπως και τα άλλα θεσμικά όργανα, προβαίνουμε σε μειώσεις κατά 5% συνολικά του προσωπικού μας. Αυτό σημαίνει ότι αν πρόκειται να γίνουν ακόμη νέα πράγματα θα πρέπει να φανούμε καινοτόμοι και ως διοίκηση και ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ταυτόχρονα να μπορούμε να εντοπίζουμε ανα πάσα στιγμή ποια καθήκοντα δεν επιθυμούμε πλέον να εκτελούμε ή ποια καθήκοντα ενδεχομένω είναι ξεπερασμένα. Και γι' αυτό το λόγο άλλωστε η μέχρι τώρα, ο μέχρι τώρα προϋπολογισμός επεγράφεται Save and Innovate και από το 2012 που είναι το έτος προπολογισμού το οποίο συζητούμε τώρα, έχουμε κοινή ομάδα εργασίας προεδρίου και Επιτροπής Προϋπολογισμών, όπου προσπαθούμε αφενός να στηρίξουμε τον απαραίτητο εξυγχρονισμό, αφετέρου να μειώσουμε κάποιες δαπάνες. Έχουμε εντοπίσει τέσσερις τομείς όπου θα επιβάλλουμε τέτοια μέτρα στην τεχνογνωσία με νέα γενική διεύθυνση επιστημονικής υπηρεσίας, επίσης στον τομέα σκρούτινη, έλεγχος, που γίνεται όλο και πιο σημαντικός και με την χρέωση των κρατών μελών, με την κρίση χρέους δηλαδή. Εκεί έχει προσληφθεί και προσωπικό. Στον τομέα της ε, διοικητικής μέρημνας, δηλαδή των, ε, των logistics, και για τα εστιατόρια αλλά και για τα γραφεία και εκεί έχουν γίνει μειώσεις και στον τομέα της στήριξης του έργου των Ευρωβουλευτών. Έχουμε λοιπόν εντοπίσει μίσο που μπορούν να γίνουν εξοικονομήσεις. Ήδη έχουν γίνει εξοικονομήσεις στον τομέα της διερμηνίας αλλά και της μεταφράσεως. Έχουμε, έχουμε μειώσει σημαντικά τι θέσεις προσωπικού αλλά έχουμε προβεί και σε βελτιωμένη οργάνωση των υπηρεσιών μείωση της χρήσεως χαρτιού, συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες, μίλησε και το ελεγκτικό συνέδριο για Streamline, το σύστημα Streamline να αντικατασταθεί από το C-Spec 2 και το Streamline να μην παραμείνει πλέον ως σύστημα μεταβίβαση δεδομένων. Για το 2012, λοιπόν, σημαντικό έτος προκλήσεων και για την εκ νέου ανακαίνιση μάλλον του κτηρίου Conrad Adenauer την οποία ανακαίνιση, στην οποία ανακαίνιση έχουμε προβεί μόνοι μας έως τώρα και από τις αρχές του έτους 2012 έχουμε καταθέσει προτάσεις για εργασίες κατασκευών οι οποίες όμως ήταν 13% άνω του ορίου που είχαμε ορίσει και γι' αυτό τις απορρίψαμε και ζητήσαμε νέες προτάσεις και έχουμε βεβαίως την πλήρη συνεργασία της Λουξεμβουργικής Κυβερνήσεως η οποία έδειξε υποδειγματική στάση, οφείλω να το ομολογήσω αυτό και οι προτάσεις τις οποίες έχουμε λάβει οδηγούν εν τέλει στο ότι μπορούμε να παραμείνουμε κάτω του προβλεπόμενου πλαισίου δαπανών για την ανακαίνιση του κτηρίου Αντενάουρ. Σας έχω ενημερώσει και για τα προβλήματα του ημικυκλίου εδώ στις Βρυξέλλες. Αφενός υπήρξε βεβαίως το πρόβλημα που είναι γνωστό, από την άλλη μεριά όμως η αναθεωρημένη μας πολιτική για την συντήρηση των κτηρίων μας επέτρεψε να εντοπίσουμε το πρόβλημα πριν να συμβεί μεγαλύτερη στατική ζημία είτε στο κτίριο ή ζημία σε βάρος κάποιων προσώπων μέσα στο ίδιο το κτίριο. Άρα η πολιτική μας επενδύσεων στην συντήρηση των κτηρίων, την οποία στήριξε άλλωστε η Επιτροπή ε, Προϋπολογισμών, αποδίδει αποτελέσματα. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι πάλι από το 2012 έχουμε βαθμιδών προχωρήσει σε νέα έννοια, σε νέο κόνσεπτ του cost accounting που όπως είπα γίνεται βαθμιδών και όπου σταδιακά θα μας οδηγήσει σε μια πολύ πιο συστηματική ανάλυση των δομών κόστους μας και θα μας επιτρέψει επίσης να μπορέσουμε να κάνουμε τις απαραίτητες μετακινήσεις κονδυλίων μέσα στον ίδιο τον προϋπολογισμό μας. Ευχαριστώ πολύ. Ο πρόεδρος Τόιρερ, ευχαριστώ πολύ. Εδώ αρχίζει βεβαίως η συζήτηση. Ο εισηγητής μας είναι ο κύριος Ήβαν και πρώτος θα, λάβει το λόγο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Βέρλε. Συνεργαστήκαμε πολύ επικοδομητικά. Σας ευχαριστώ λοιπόν για τη συνεργασία αυτή και πιστεύω θα συνεχιστεί και στο μέλλον. Συνεργαστήκαμε πολύ καλά επίσης και με τους Γενικούς Διευθυντές. Είχαμε πολύ επικοδομητικές συναντήσεις, ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες. Θα ήθελα λοιπόν να σας συγχαρώ κύριε Γενική Γραμματέα, διότι καταφέρατε να ενισχύσετε το ρόλο του εσωτερικού ελεγκτή. Ο εσωτερικός ελεγκτής είναι πλέον πολύ πιο παρόν, συμμετέχει πολύ περισσότερο στις διάφορες δραστηριότητες του Κοινοβουλίου και εγώ συνεργάστηκα μαζί του. Είχα τη δυνατότητα να συζητήσω μαζί του και να ευχαριστήσω και τον Αντιπρόεδρο κύριο Τζάνι Πιτέλα γιατί έχει πολύ καλές επαφές με την Επιτροπή μας, Ελέγχο του προπολογισμού, είναι αρμόδιος άλλωστε για τον προπολογισμό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα ήθελα να τον ευχαριστήσω και αυτόν μόνο ότι απουσιάζει σήμερα. Να ευχαριστήσω επίσης γενικότερα τη διοίκηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διότι καταφέραμε να αντιμετωπίσουμε περίπου, μάλλον υποβάλαμε 140 ερωτήσεις και λάβαμε πολύ σαφείς ξεκάθαρες απαντήσεις. Όπως είχα τη δυνατότητα να το πω και παλαιότερα, διανύουμε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Θα ψηφίσουμε την έκθεση αυτή και στη συνέχεια θα περάσουμε στην προεκλογική περίοδο. Υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι ήδη βρίσκονται στα πλαίσια μιας προεκλογικής εκστρατείας και ξέρετε ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τα δημοσιονομικά ζητήματα και πολλές φορές ασχολούνται ως προς αυτό με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το 2012 ήταν θα έλεγα μια θετική χρονιά από δημοσιονομικής πλευράς για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, βελτιώθηκαν οι παρεχόμενε υπηρεσίε και μειώθηκε το κόστο παράλληλα. Βέβαια έχουμε και μία αξιολόγηση, τον έλεγχο από τον εξωτερικό ελεκτή, από το ελεκτικό συνέδριο. Η αξιολόγηση αυτή είναι θετική όπως ακούσαμε. Θα ήθελα όμως να αναφερθώ και στην εσωτερική αξιολόγηση που έλαβε χώρα. Δεν θα ήθελα να μακρηγορήσω. Θα μπορούσα πάντως εν συντομία να αναφερθώ σε κάποιες πτυχές του ελέγχου αυτού. ιδίως όσον αφορά την αναδιάρθρωση της DigiTrad, IMCO και COM. Γίνανε για τις τρεις αυτές γενικές διευθύνσεις κάποιες τροποποιήσεις, κάποιες αλλαγές που τις κατέστησαν πιο αποτελεσματικές, ενώ παράλληλα μειώθηκε το κόστος στο οποίο αντιστοιχούσαν οι τρεις αυτές γενικές διευθύνσεις. Τι ακριβώς λοιπόν έγινε σε αυτές τις γενικές διευθύνσεις, ποιο είναι το ποσό το οποίο καταφέραμε να εξοικονομήσουμε. Πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι που διαρωτώνται αν η Ολομέλεια του Απριλίου τελικά θα μπορέσει να λάβει χώρα εδώ, στο Μικύκλιο των Βρυξελών. Ολοκληρώνω στο σημείο αυτό. Yeah. θα δώσω τον λόγο στον εσωτερικό ελεγκτή του Ευρωπαϊκού ε, Κοινοβουλίου, ο κύριο Ρόμπερτ Κάλβιν. Πού βρίσκεστε, αγαπητοί κύριοι. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Πρώτα πρώτα, πρόεδρε, να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μας δίνετε να σας παρουσιάσουμε για το 2020 2012, συγγνώμη, την ε, ετήσια έκθεση που δίνει το αποτέλεσμα των εσωτερικών ελέγχων κατά την χρήση εκείνη. Επίση, θα πρέπει να σα υπενθυμίσω ότι εκεί που επισημαίνουμε κάποια προβλήματα προτείνουμε κάποιες δράσεις υπό τη μορφή των συστάσεων. Και έτσι υπάρχει συνεχής διάλογος, διαβούλευση με τις υπηρεσίες και προσπαθούμε να πετύχουμε κάποια συμφωνία. Το 2012 Κάναμε τον οικονομικό έλεγχο και έχουμε το κάθε πρόγραμμα το οποίο προκύπτει από την αξιολόγηση κινδύνων. Ο σκοπός είναι η υπηρεσία μας να μπορεί να δώσει προτεραιότητες για το πού θα, πώς θα κατανείμει τέλο πάντων το, τους που έχουμε εκεί που επιβάλλεται. Το 2012 στην προσοχή μας σε μια νέα προσέγγιση ούτως ώστε να δοθεί κάποια συνέχεια τον είχαμε προηγουμένω. πριν είχαμε την εξέδεση κάθε δράση όταν χθε εξέπνιαν με την καινούργια προσέγγιση προσπαθούμε δύο φορές το χρόνο να ελέγξουμε τι γίνεται και να, και να τις επικυρώσουμε σε σχέση και με τις προηγούμενες εκθέσεις και έτσι το 2013 ε, καλύψαμε 153 από 21 προηγούμενες εκθέσεις. 80 από αυτές τις κλείσαμε και οι υπόλοιπες 72 θα ε, πρόκειται να εκκρεμούν για την έγκριση. Και είχαμε 30 δράσεις που θεωρήσαμε ότι θα έπρεπε να αξιολογηθούν περαιτέρω όσον αφορά τον κίνδυνο που ενέχουν. Το 2012 επίσης είδαμε το πόσε είναι οι δράσεις οι οποίες ε, διαπνύονται από κάποιο ιδιαίτερο κίνδυνο, από 8 ήταν 2 είπαμε και επίσης από την επιμελητία θεωρήσαμε ότι στην διαδικασία των προμηθειών είχαμε βελτιώσεις και έγιναν σημαντικά διαβήματα όσον αφορά ε, τα, της και επίσης ε, κλείσαμε κάποιες δράσεις όσον αφορά το πλαίσιο των εσωτερικών ελέγχων και έτσι η διαχείριση των επιδόσεων ήταν ένα σημαντικό θέμα. Οπότε και έτσι έμεινε ε, ανοιχτέ κάποιες δράσεις ε, παρά το ότι μειώθηκε ο κίνδυνος που αξιολογήθηκε όσον αφορά τα πολιτικά κόμματα και τα ιδρύματα. Τέσσερις από τις 36, ε, έμειναν ανοιχτέ και ακόμα θα πρέπει να γίνει η αξιολόγησή τους. Είχαμε δαπάνες από κάποια ταμεία Είχαμε κάποια σημεία περιμερία οπότε είπαμε ότι θα έχουμε εφαρμοστικά μέτρα σύμφωνα με τον νέο δημιουργικό κανονισμό και το νέο σύστημα χρηματοδότησης. Για να δούμε τώρα τι άλλο έγινε το 2012. Ο ελεγχο ήταν αντικείμενο του πέμπτου ελέγχου που έγινε. Και σύμφωνα αυτόν τον έλεγχο καταλήξαμε ότι γενικά οι δράσεις που ελέγχθηκαν σε όλες τις γενικές διευθύνσεις προκύπτει ότι όλα έγιναν σύμφωνα με τους κανόνες της στρατηγικής που είχε χαραχθεί. Επίσης είδαμε ότι αναβαθμίστηκαν κάποιες διαδικασίες σε σχέση με την μετρίου μεγέθους εκθέσεις σε κίνδυνο. Οπότε έτσι είπαμε ότι κάποιες από αυτές τις δαπάνες θα, δεν θα καταβληθούν μέχρι το τέλος των συμβάσεων πρόσληψης αυτών των συνεργατών. Είπαμε ότι μετά τις εκλογές του 2014 πρόκειται να προσληφθούν κάποιοι άλλοι συνεργάτες και γι' αυτό και έχουμε κάποιο πρόγραμμα δράσης με τις αρμόδιες γενικές διευθύνσεις και το 2012 κάτι άλλο που έγινε είχαμε τον έλεγχο ε, των κάποιων ε, λογιστικών. Και έτσι είπαμε ότι αυτά συνάδουν προς τον δημοσιονομικό οργανισμό και τα όσα ισχύουν στα άλλα θεσμικά όργανα. Θα έπρεπε να δούμε κατά πόσο αυτές οι διαδικασίες είναι ε, αποτελεσματικές και αν υπάρχει η σωστή πλαισίωση από την πληροφορία και αυτό είπαμε ότι έχουμε κάποιες κάποια έκθεση σε κινδύνους. Όσον αφορά τα ακίνητα, την περιουσία του Κοινοβουλίου, είπαμε ότι θα γίνει κάποια αξιολόγηση από τι λογιστικέ υπηρεσίε και θα έπρεπε επομένω τη λογιστική αυτή διαδικασία να αξιολογηθεί και αυτό να γίνει επί τη βάση της ε, πληροφορικής όπως υπάρχει σαν υποστήριξη και γι' αυτό είπαμε ότι θα πρέπει και οι συμβάσεις των συνεργατών μας να διέπονται ε, από τον δημοσιον κανονισμό. Επίσης, το 2012 είχαμε και κάποιες διαδικασίες παροχής συμβουλών και αυτό έχει να κάνει και με κάποιο πρωτόκολλο του διαδικτύου οπότε συμφωνήσαμε με τον πάροχο αυτών των υπηρεσιών διαδικτύου. Έτσι θα έπρεπε να δούμε τα εξή ζητήματα. Πρώτα πρώτα. Το 2006-2007 είχαμε 5.000 ε, τηλέφωνα. Και επίσης είπαμε ότι δεν υπήρχε διαφάνεια στι αρχές αποφάσεις να συνεχίσουμε με αυτό το πρόγραμμα γιατί υπήρχε συγκεκριμένο κατασκευαστή τηλεφώνων που θα έπρεπε να εξεταστεί η σύμβασή του. Καταλήξαμε σε 23.000 χρήστες αυτών των υπηρεσιών. Αυτά τα ζητήματα πέρασαν από τον ιστορικό έλεγχο και κάναμε κάποιες συστάσεις προς τη Γενική Διεύθυνση της Πληροφορικής, της ITEC. έγινε ανταλλαγή παλαιότερων συσκευών με νέες. Είχαμε κάποιες μελέτες για να πάμε προς νέους προμηθευτές και είπαμε ότι θα πρέπει να αλλάξει ο τρόπος λήψης των αποφάσεων, να βελτιωθεί. Πολιτική κτηρίων. Και εδώ ασκήσαμε έλεγχο, να δούμε τι κίνδυνοι υπάρχουν. Και 23 Τρίτου του 10 αποφάσισε το Προεδρείο να υπάρξει κάποια πολιτική διδακτήρια και είπαμε ότι έγιναν βήματα πρόοδου όσον αφορά την πολιτική αυτή των κτηρίων του Κοινοβουλίου. Πιστοποίηση, ασφάλεια και έχουμε κάποιους εξωτερικούς αξιολογητές στον τομέα των κτηρίων. Νέα διαδικασία, αναθεωρημένη, πιο σύντομη έλεγχη σύμφωνα με τις προτεραιότητες που έχουμε. Έχουμε προγράμματα δράσης σε αυτόν τον τομέα. Μετά είπαμε ότι θα πρέπει να υπάρξει κάποια διαδικασία ελέγχων για τους κινδύνους, διοίκηση, διαχείριση, τι γίνεται με τα πάνελ σύμφωνα με τις άριστες πρακτικές και την χρηστή διακυβέρνηση. Κατόπιν έχουμε τα συμπεράσματα του εσωτερικού ελέγχου, κυρίως όσον αφορά την διαδικασία εποπτείας, οπότε γενικά διαπιστώθηκε βελτίωση και βελτίωση της παρακολούθησης των κινδύνων σε κάθε υπηρεσία, σε κάθε τομέα. Άρα το 2013 θα σε κάλυψη 75% των όσων θέλαμε. Επίσης υπάρχουν στοιχεία προόδου για τους συνεργάτες μας σε σχέση με τον προηγούμενο ιστορικό έλεγχο της προηγούμενης χρήσης. Και είπαμε ότι σύστημα 2011 δεν έχουμε επιδείνωση όσον αφορά την αμεροληψία και το των ελέγχων. Ε, πρέπει να ευχαριστήσω όλους όσους ελέγξαν το 2012 για τις συνεργασία τους και ευχαριστώ. thank you very... Ο Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ και Colin, όχι μόνο για την έκθεση που παρουσιάσατε αλλά και για το έργο που είναι σημαντικό, το έργο σας. Βεβαίω, πάντα των ελεγκτών είναι πολύ σημαντικό, ίσως οι ίδιοι να μην είναι οι πιο αγαπητοί άνθρωποι, αλλά είμαι πεισμένος ότι το έργο σα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και τώρα επιτρέψτε μου να θέσω ε, την έκθεση υποσυζήτηση και βεβαίω πρώτη η κυρία Πορτίθ Βιλέγια από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε, καλώς όρισατε κυρία Γενικέ. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε να μας δείτε και να διευθυνήσουμε κάποια ζητήματα. Ευχαριστούμε και τους εκπροσώπους του συνεδρίου, τον εσωτερικό έλεγχο και τους συναδέλφους βέβαια. Έχω κάποιες ερωτήσεις. Αν και βέβαια ε, ενώ έχουν υπάρξει σήμερα με το ερωτηματολόγιο κάποιες απαντήσεις δεν έχω καταλάβει πολύ καλά. Τι γίνεται με το ημικύκλιο και την σύνοδο του Απριλίου. Μας τα είπατε. Αλλά ξέρουμε τελικά πόσο θα κοστίσουν οι επισκευέ. Άλλαξε κάτι σε σχέση με αυτά που ξέρουμε, αυτά που μας έχετε πει. Τι αλλάζει όσον αφορά πάντων τον προπολογισμό, όσον αφορά τον προγραμματισμό, την διαχείριση, τις προμήθειε, όλα αυτά. Αυτό μα απασχολεί τι πρωτοβουλίες, τι μηχανισμοί ελέγχου έχουν ενεργοποιηθεί ούτως ώστε να εξηγιάνουμε την κατάσταση εκεί που, έπασχε, ε, εκεί που έπασχαν οι, οι, οι σχετικές διαδικασίες Ε, τι τι άλλε ε, ε, διαπραγματεύσει έγιναν για κάποιε εξαιρετικέ καταστάσει. Επίση, για πετε μα, έχετε ενεργοποιήσει κάποιο είδου διαδικασία ενεργοποίηση από κάποιον ανεξάρτητο όσον αφορά τι συμβάσει για, για, με, με κάποιου εξωτερικέ εταιρείε. Επίση, Καλώ ήρθατε και εσωτερική ελεγκτά. Πέστε μα όμω, τι γίνεται όσον αφορά τα συμπεράσματα του προγράμματο δράση για τη βελτίωση των υπηρεσιών εσωτερικού οικονομικού ελέγχου για όσα όφυλαν να γίνουν στο τέλο του 2012 για όσα αποφασίστηκαν τότε. Επίση, εν κατακλείδη, έχουμε την έκθεση αξιολόγηση για ε, το κόστο σε σχέση την αποτελεσματικότητα του, της ε, Europa TV. Τι γίνεται, το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό. Ευχαριστώ. Ας ακούσουμε πρώτα ώρες τις ερωτήσεις και ακολουθεί ο κύριος Μάρτιν. Ευχαριστώ. Έχω θέσει πολλές ερωτήσεις όπως θα είδατε στον κατάλογο που υπέβαλα και θα ήθελα τώρα να επανέλθω σε ορισμένες που δεν απαντήθηκαν. Και θα ήθελα να ρωτήσω εσάς κύριε Γενική Γραμματεύ να σας παρακαλέσω αν είναι δυνατό να με διαβεβαιώσετε ότι θα μου απαντήσετε για, τα συγκεκριμένα, για το συγκεκριμένο κόστος των πτήσεων των Ευρωβουλευτών για το 2012. Οι τρεις ακριβότερες, τα πανηρότερες δηλαδή αποστολές, επίσης το κόστος των συνεργατών του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες ερωτήσεις ο ίδιος είπατε και όντως θεωρώ ότι είναι θετική εξέλιξη ότι το κόστος των μεταφράσεων έχει μειωθεί. Όμως έχω κάνει συγκεκριμένες ερωτήσεις σχετικά που δεν μου απαντήσατε. Το ίδιο για τις πρόορες συνταξιοδοτήσεις ορισμένων υπαλλήλων του Κοινοβουλίου, καθώς επίσης για το κόστος καθαρισμού των κτηρίων του Κοινοβουλίου. Θα ήθελα λοιπόν να λάβω απαντήσεις για τις ερωτήσεις αυτές. Και επειδή δεν είναι εύκολο να σας συναντήσω ή να μιλήσω μαζί σας ως Ευρωβουλευτής, τονίζω ότι σας έχω αποστείλει και δύο επιστολές. Η μία αναφέρεται στη συγκεκριμένη στάση των υπαλλήλων της ασφαλείας που πληρώνονται από χρήμα των φορολογμένων και οι οποίοι με παρακολουθούν επί ώρες και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω λοιπόν και εκεί τις ερωτήσεις αυτές και ότι ακόμα αναμένω τις απαντήσεις σας. Ευχαριστώ. Ακολουθεί ο κύριος Μιλντερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εάν δεν κάνω λάθος, οι επισκευές για την στέγη, για την οροφή δηλαδή του ημικυκλίου στο Στρασβούργο καλύπτεται από τις εγγυήσεις που είχε δώσει ο κατασκευαστής. Τώρα στο ημικύκλιο εδώ της Βρυξέλλες θα πληρώσουμε εμείς, έτσι δεν είναι. Επίσης, οι πληρωμές που γίνεται τώρα ευθυγραμμίζονται με όσα αναμέναμε. Ευχαριστώ κυρία Γκρέσλε. Ευχαριστώ. Μία παράκληση ο εσωτερικός ελεγκτής να μας διαβιβάσει την παρουσίασή του, γιατί διάβασε με τέτοια ταχύτητα που δεν μπόρεσα να παρακολουθήσω. Δεύτερο, για την οροφή στις Βρυξέλλες με κόστος επισκευών της τάξης των 2 εκατομμυρίων ευρώ. Υπάρχει κάποια δική μας αντίδραση στο νομικό επίπεδο, μπορούμε να ζητήσουμε κάποια αποζημίωση από τον κατασκευαστή. Θα ήθελα αυτές τις πληροφορίες. Επίσης, το έλλειμμα 207 εκατομμυρίων του εθελοντικού συστήματος συντάξεων των Ευρωβουλευτών. Μπορεί αυτό το Ταμείο να επιβιώσει. Τι γίνεται. Από ποια στιγμή και μετά τα πράγματα θα, είναι, θα φτάσουν στο απροχώρητο. Έχω και μια άλλη υπόθεση που το ποσόν δεν είναι ίσως τόσο σημαντικό, αλλά τίθεται θέμα αρχής. Το Κοινοβούλιο έδωσε μια επιδότηση, ένα grant, κάτι το οποίο βρίσκω αρκετά ασυνήθιστο, σε μια βουλγαρική φύρμα, η οποία εν τω μεταξύ αποδείχτηκε ότι ανήκει στον, ε, στην σύζυγο ενός αναπληρωτού προέδρου της, ε, του Σοσιαλιστικού Κόμματος της τάξης 60.000 ευρώ. Εγώ βρίσκω ότι πρόκειται για καθαρή σύγκρουση συμφερόντων. Γιατί δεν ακυρώνεται η πληρωμή αυτή όταν ένας εντελοδόχος λαμβάνει από το Κοινοβούλιο ένα ποσό και όταν λέει ο κανονισμός καθαρά ότι χρειάζεται, οφείλει να δοθεί στην περίπτωση αυτή ένορκη δήλωση ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Εγώ ε, ασχολήθηκα λίγο με την υπόθεση αυτής της εταιρεία και βλέπω ότι η εταιρεία, αυτή εμπλέκεται σε ένα σκάνδαλο στην Αυστρία. Η βουλγαρική κυβέρνηση έδωσε 1,5 εκατομμύρια ευρώ σε κάποιον αυστριακό έγκερ ο οποίος ασχολείται με δημόσιες σχέσεις και πάλι εκεί εμπλέκεται αυτή η εταιρεία τους, της συζύγου του ε, αντιπρόεδρου του Σοσιαλιστικού Κόμματος στη Βουλγαρία. Αν να τέτοια πράγματα στη Γερμανία θα ξεσπάσει μέγα σκάνδαλο. Υπάρχει και εμπλοκή μιας βελγικής εταιρείας. Και αν εξετάσει κανείς τον ισολογισμό που προέρχεται το 2008, βλέπει κανείς μια έλλειψη, ένα έλλειμμα μάλλον, της τάξης των 84.000 ευρώ στον ισολογισμό της εταιρείας αυτής. Γι' αυτό και διαρωτώ Αυτές οι 60.000 ευρώ της επιδοτήσεως πώς είναι δυνατόν να έγιναν. Θα ήθελα να μπορέσουμε να ξεφορτωθούμε την εταιρεία αυτή. Εδώ μου γράφουν από τη μισή Ευρώπη για την υπόθεση αυτή. Όχι από Βουλγάρους, από πολλούς άλλους που μου λένε ότι δεν είναι δυνατόν να κάνετε τέτοια πράγματα, να εγκρίνετε τέτοια πράγματα. Αυτά, ευχαριστώ. Όντω οι ερωτήσει σα είναι σημαντικέ. Μια στιγμή να δω τώρα, λέει ο πρόεδρο Νομίζω ότι ακολουθεί η κυρία Σέντερ, Αγιάλα Σέντερ. Αν δεν έχω δει κάποιον, παρακαλώ να μου το θυμίσει. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για τον κύριο Βέλε που ήρθε. Θα ήθελα να τον ρωτήσω. Μήπως θα μπορούσατε να μας εξηγήσετε τα βασικά σημεία της αναδιοργάνωσης της ε, γραμματείας μας εν ώψη των όσων θα γίνουν. νέε αρμοδιότητε, ό,τι μπορείτε να μα εξηγήσετε. Επίση, πρόσφατα είχαμε αυτή την επίθεση απ' έξω. όσον αφορά την υπηρεσία πληροφορική του Κοινοβουλίου. Εμεί προσπαθήσαμε να κάνουμε ό,τι και να λάβουμε τη μέτρα μπορούσαμε. Όμω, το αποτέλεσμα είναι τώρα οι επισκέπτες δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στο ασύρματο δίκτυο του Κοινοβουλίου. Το έχουμε ήδη συζητήσει αυτό. Για πέστε μας. Πώς θα αντιμετωπίσουμε τέτοιες περιπτώσεις, τέτοιες εξωτερικές επιθέσεις. Αυτά ε, όλο ένα και εντείνονται ως φαινόμενα αυτούς τους hackers. Και το θέμα δεν είναι ότι εδώ έχουμε τίποτα τρομερά, απόρριτα και κρατικά, αλλά θέλουν να κατασκοπεύουν τις διαπραγματεύσεις όσα λέμε. Έχει βελτιωθεί πάρα πολύ σημαντικά οι υπηρεσίε της βιβλιοθήκης μας, αυτά τα, τα δελτία, τα ενημερωτικά, όλα αυτά για την ε, προσεχή προεκλογική στα θα είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Ήταν πάρα πολύ σωστή εκείνη η ιδέα του Προεδρείου να υπάρχει μια τέτοια υπηρεσία με αυτή τη μορφή. Νομίζω ότι λειτουργεί καλά. Δεν έχουν ενημερωθεί όλοι βέβαια για την ύπαρξη και την επίδοση αυτή τη βιβλιοθήκη, αλλά όσοι ξέρουμε, ξέρουμε ότι είναι μια χαρά. Äh, Ευχαριστώ. Δεν έχω άλλου εγγεγραμμένου για την ώρα, ώστε δίνω το λόγο σε εσά κύριε Γενική Γραμματεύ για να απαντήσετε. Μάλιστα, σας ευχαριστώ. Πρώτα για τις ερωτήσεις του εισηγητού. Υπήρξαν όμως και ορισμένες επικαλύψεις και με άλλους, για παράδειγμα για το θέμα της οροφής του ημικυκλίου, όπου θα προσπαθήσω να τις συνοψίσω. Πρώτα λοιπόν για το ημικύκλιο. Αρχικά θεωρήσαμε ότι η επισκευή θα έφτανε έως 3 εκατομμύρια ευρώ Τώρα φτάνουμε στα 2, ίσως 2,3 εκατομμύρια και νομίζω ότι θα αρκέσουν τα χρήματα αυτά. Έχουν σχεδιαστεί οι εργασίες ήδη πριν από τις διακοπές των Χριστουγέννων. Ε, είχαμε μια καθυστέρηση δύο εβδομάδων, αρχές Δεκεμβρίου. Η εταιρεία μας έχει διαβεβαιώσει ότι θα εργάζεται 7 ημέρες την εβδομάδα, χωρίς καμία διακοπή λοιπόν. Έχει έλθει η νέα δομή, άρα έχει ήδη εγκατασταθεί η νέα δομή και στηρίζει την οροφή, μένει βέβαια η έγκριση από τις αρμόδιες αρχές, η οποία θα γίνει τις ημέρες αυτές. Έχει λοιπόν εγκατασταθεί η νέα δομή, αλλά θα πρέπει, όπως είπα, να γίνει επιθεώρηση και έγκριση από τις αρμόδιες αρχές. Εφόσον γίνει αυτό επιτυχώς, θεωρώ ότι θα παραμείνουμε μέσα στο χρονοδιάγραμμα, Άρα, όσοι έχουν τα πράγματα για την ώρα, δεν φαίνεται να υπάρχει ο φόβος η μήνυ ολομέλεια του Απριλίου να μην μπορέσει να διεξαχθεί εδώ. Παρόλο λοιπόν που το εγχείρημα ήταν πολύ δυσχερές γιατί η οροφή χρειάστηκε μάλιστα να υψωθεί λίγο για την ώρα θεωρούμε ότι βρισκόμαστε μέσα στο χρονοδιάγραμμα και υποθέτω λοιπόν όπως είπα ότι η μήνυ ολομέλεια του Απριλίου θα μπορέσει να διεξαχθεί σύμφωνα με το πρόγραμμα τον προγραμματισμό. Για τα νομικά θέματα τα οποία θίξατε ορισμένοι εξημών, στον χώρο του ημικυκλίου των Βρυξελών είμαστε πλέον εκτός του χρόνου εγγύησεως της δεκαετίας. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να εγείρουμε απαιτήσει διότι όπως είπα έχει παρέλθει η δεκαετής περίοδο εγγύσεως. Επιπροσθέτως, ο κατασκευαστής της οροφής έχει σεβαστεί στην κατασκευή τους κανόνες που ίσχυαν τότε. Το, το πρόβλημα είναι ότι επρόκειτο για μια νέου είδους ξύλινη κατασκευή η οποία και ό,τι μάλιστα συμπληρώνω μετά ναι. από την κατασκευή της στέγης αυτής, τροποποιήθηκαν οι κανονισμοί και μάλιστα κατ' επανάληψη. Όμως, ο αρχικός κατασκευαστής δεν βαρύνεται, διότι είχε κατασκευάσει την δομή αυτή σύμφωνα με τους τότε ισχύοντες κανονισμούς. Άρα εν τέλει εδώ δεν έχουμε καμία δυνατότητα να ζητήσουμε αποζημίωση. Ο εισηγητής μου ζήτησε επίσης πληροφορίες για τις διάφορες αναδιαρθρώσεις εντός του Κοινοβουλίου που έχουν επηρεάσει πλήονες γενικές διευθύνσεις, Γενική Διεύθυνση Μεταφράσεων για παράδειγμα, από τις οποίες μετακινήσαμε 100 θέσεις του οργανογράμματος σε άλλες υπηρεσίες για την πολιτική στήριξη, για παράδειγμα, των βουλευτών. Επίσης σημειώθηκαν οι δαπάνες για εξωτερικές μεταφράσεις κατά 10 εκατομμύρια ευρώ. Έχουν γίνει σημαντικές εξοικονομήσεις λοιπόν εν τέλει στην υπηρεσία μεταφράσεων. Η συνέπεια είναι ότι η καθαρή παραγωγικότητα ανασυνεργάτη έχει ανέλθει και πέρσι το 2013 έχουμε φτάσει στις 7,7 σελίδες ανασυνεργάτη πάρα πολύ υψηλή τιμή, όχι όμως με την έννοια ότι ορισμένοι εργάζονται περισσότερο, αλλά ότι τώρα βαρύνονται με τον ίδιο περίπου φόρτο εργασίας, εργασίας όλοι λίγο πολύ οι μεταφραστές. Ή, βρισκόμασταν παλαιότερα σε μια κατάσταση όπου ορισμένα μεταφραστικά τμήματα είχαν λιγότερο φόρτο εργασίας από άλλα. Ε, πρόκειται για μια έλλειψη ισορροπίας η οποία εν τέλει μπόρεσε να αρθεί. Έτσι λοιπόν σήμερα η απόδοση αναμεταφραστεί αποκλίνει ελάχιστα ανάμεσα στα διάφορα μεταφραστικά τμήματα. Το πλεονασματικό αυτό προσωπικό μπόρεσε να διατεθεί σε άλλες υπηρεσίες, για παράδειγμα για την στελέχωση του οίκου της Ευρωπαϊκής Ιστορίας, για την ε, ε, υπηρεσία που ασχολείται με το follow-up. υπηρεσίες που στελεχώθηκαν χωρίς αύξηση του οργανογράμματος. Εδώ έχω να σας δώσω και ένα πρόσθετο αριθμό. Τα τελευταία 10 χρόνια η παραγωγή της μεταφράσεως από 1 εκατομμύριο σελίδες τον χρόνο έχει ανέλθει σε 2,5 εκατομμύρια τον χρόνο μέσα σε 10 χρόνια. Και αυτό παρόλο που ο συνολικός αριθμός προσωπικού εν τέλει μετά από τις αλλαγές που εξήγησα δεν έχει ανέλθει σχεδόν καθόλου και παρόλο που μειώθηκαν οι δαπάνες εξωτερικών μεταφράσεων. Αυτό κατέστη δυνατόν λόγω δύο παραγόντων. Αφενός χρήση σύγχρονων τεχνολογιών περίπου το 40% τώρα προμεταφράζεται διότι παρόμοια κείμενα έχουν μεταφραστεί ήδη και επομένως δεν χρειάζεται να ξαναμεταφραστούν από την αρχή Δεύτερο, η αύξηση της παραγωγικότητας που επετεύθη, δηλαδή πρόκειται για πραγματική έκρηξη μεταφραστικού έργου, που ευτυχώς όμως δεν συνοδεύτηκε από έκρηξη του κόστους. Και όπως είπα, ιδίως χάρη στην σύγχρονη τεχνολογία, αλλά και με καλύτερη κατανομή του προσωπικού μέσα στα πλαίσια της Γενικής Διεύθυνσης. Τώρα, για τη Γενική Διεύθυνση Διερμηνίας. Πάλι εκεί μπορέσαμε να μετακινήσουμε από αυτή την Γενική Διεύθυνση 40 περίπου θέσεις, οργανικές θέσεις, κάτι που οδήγησε σε μείωση θέσεων σε ορισμένα τμήματα τα οποία δεν είχαν ιδιαίτερο φόρτο εργασίας και μπορέσαμε να οδηγηθούμε σε εξοικονόμηση περίπου 15 εκατομμυρίων ευρώ τον χρόνο. Αυτά δεν είναι εφάπαξ μόνο εξοικονομήσεις, είναι διαρθρωτικές εξοικονομήσεις σε βάθος χρόνου. Επομένως μπορούμε με τον τρόπο αυτό να προβούμε σε καλύτερο σχεδιασμό. Επίσης οι κοινοβουλευτικές επιτροπές συνεδριάζουν πλέον και Δευτέρα απόγευμα και Πέμπτη, όχι όλες πλέον Τρίτη, Τετάρτη αποστολές αντιπροσωπιών γίνονται όλο και περισσότερο στις λεγόμενες γαλάζιες εβδομάδες, κάτι το οποίο βεβαίως σημαίνει κάποια πειθαρχία από πλευράς των Ευρωβουλευτών, από την άλλη μεριά όμως εξοικονομούμε σημαντικό κόστος σε προσωπικό. Έχουμε επίσης μπορέσει να βελτιώσουμε το σχεδιασμό της ε, Ολομέλειας του Στρασβουρού και κυρίως τις νυκτερινές συνεδριάσεις, άρα και στην διερμηνία και στη μετάφραση μπορέσαμε να κάνουμε σημαντικές εξοικονομήσεις και σε ό,τι αφορά την χρήση εξωτερικών πόρων αλλά και στην χρήση των, του προσωπικού μας και μάλιστα σε ένα χρόνο όπου βρισκόμαστε προς το τέλος πλέον της κοινοβουλευτική θητείας και επομένω ο φόρτος εργασίας αυξάνεται. Η αναδιάρθρωση και στην Γενική Διεύθυνση Εξωτερικών Πολιτικών έχουμε εκεί την ε, νέα υπηρεσία που ωστόσο ήταν ουδέτερη από άποψη ε, προσωπικού, δεν χρειάστηκαν δηλαδή να γίνουν εξοικονομήσεις. Έχουν γίνει και περιφερειακές υπηρεσίες. Βέβαια ένα συνεργάτης μπορεί να είναι πολύ αποδοτικότερος ε, εφόσον δεν είναι αρμόδιος για μια χώρα στη Λατινική Αμερική, στην Αφρική και στην Ασία, αλλά συγκεντρώνει την προσοχή του σε μία περιοχή του κόσμου. Και αυτό λοιπόν σημαίνει μείωση του κόστου. Στη Γενική Διεύθυνση ΙΝΛΟ, δηλαδή τα κτίρια, πρόκειται για ένα έργο το οποίο ξεκινήσαμε ήδη το 2009 με την δημιουργία ειδική διεύθυνση για την συντήρηση των κτίριων, κάτι το οποίο τότε κόστησε με χρήματα, γιατί δημιουργήσαμε 47 έξτρα οργανικές θέσεις και είχαμε εγκρίνει και σχετικά κονδύλια, στο μεταξύ όμως αποδεικνύεται καλή επένδυση, διότι η εν λόγω διεύθυνση και η νέα, ο νέος κατασμερισμός έργου μπόρεσε να αποκαλύψει τις αδυναμίες του κτηρίου της Βρυξέλλες, διότι αν δεν είχαν αποκαλυφθεί οι σχετικές αδυναμίες θα είχε καταρρεύσει η οροφή και πιθανότατα με πολύ δραματικότερο τρόπο από ό,τι έγινε στο Στρασβούργο διότι γνωρίζετε ότι το κτίριο εδώ δεν χρησιμοποιείται μοναχά για ολομέλειες, αλλά και για συνεδριάσεις επιτροπών. Και μπορούμε να έχουμε εκεί μέχρι και 200 συνεργάτες οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στην ε, αίθουσα αυτή. Φαντάζεστε τι δραματικό θα ήταν, τι δραματική θα ήταν η καταστροφή, γι' αυτό θεωρώ ότι η επένδυση που κάναμε για την συντήρηση των κτηρίων με δημιουργία ειδική διεύθυνση και με τακτικές επιθεωρήσεις από εμπειρογνώμονες ήταν μια πραγματικά χρήσιμη επένδυση. Και την βρίσκω απόλυτα δικαιολογημένη. Και δεν θα βρισκόμουν εδώ μπροστά σας αν δεν είχαμε κάνει τότε αυτή την επένδυση. Στην Ίνλο ξεχωρίσαμε τους κλητήρες που είναι αρμόδιοι για την εξυπηρέτηση των αιθουσών και εκείνου που κάνουν τη μετακίνηση των ταχυδρομείων. Σε δεύτερο βήμα εξετάσαμε τον αριθμό των συνεργατών μας που μεταφέρουν έγγραφα, ταχυδρομείο κλπ. Και μπορέσαμε να τους μειώσουμε κατά το 1 τρίτο. Λογικό είναι βέβαια αυτό, διότι εν τω μεταξύ, πιστέψτε το ή όχι, παράγουμε πολύ λιγότερο χαρτί. Στα τελευταία 10 χρόνια μπορέσαμε να μειώσουμε κατά 60% τη χρήση χαρτιού στο τυπογραφείο. Και επομένω λιγότερο χαρτί χρειάζεται και να μετακινείται, να μεταφέρεται. Οι θέσει αυτέ που εξοικονομήθηκαν μπόρεσαν να τοποθετηθούν αλλού, ιδίω στο One Stop Shop των Ευρωβουλευτών, όπου προσφέρει υπηρεσίε στου Ευρωβουλευτέ και θα αρχίσει να προσφέρει τι υπηρεσίε αυτέ από αρχέ Φεβρουαρίου και εκεί μπόρεσε να στελεχωθεί η υπηρεσία αυτή χωρίς νέες, νέες θέσει. Τα μέτρα που λήφθηκαν επίσης για τη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιών ήταν κάπως πιο περιορισμένοι. Έχουμε τον οίκο της Ευρωπαϊκής Ιστορίας που εν, μέρη συγγνώμη, λειτουργεί με συμβασιούχους, κυρίως όμως με πλήρεις υπαλλήλου και αυτοί μετακινήθηκαν από άλλες υπηρεσίες, ώστε και εκεί δεν προκλήθηκε έξτρα κόστος. Ο τομέας τύπου έχει την ίδια διάθρωση όπως και άλλοι τομείς, για παράδειγμα η νομική υπηρεσία, η υπηρεσία των επιτροπών ή και οι γλωσσικές υπηρεσίες. Αυτά σχετικά με την επισκόπηση των αναδιαθρώσεων και των επιπτώσεών των. Η κυρία Ορτής έθεσε την ερώτηση σχετικά με τις έκτακτες διαδικασίες, exceptional procedures, θέμα το οποίο παρακολουθούμε εδώ και καιρό Ίσως είναι δυνατόν αυτό που είπατε πράγματι. Για το 2013 μπορώ να πω ότι οι exceptional procedures μειώθηκαν. Από 58 τον προηγούμενο χρόνο έφτασαν 45. Άρα οι τάσεις είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Εν πάση περιπτώσει παρέμειναν 45 έκτακτες διαδικασίες. Και εν πάση περιπτώσει, ξαναλέω, το έχω τονίσει άλλωστε αυτό, η διαβούλευση με το Procurement Forum είναι δυνατή, πρόκειται για συμβουλευτικό όργανο, η δε διαβούλευση μαζί του είναι υποχρεωτική και το υπενθύμησα αυτό και πάλι. Κάνατε και άλλη μια ερώτηση για την πληροφορική, δηλαδή την εξάρτησή μας από εξωτερικές εταιρείες. Εδώ το Προεδρείο απεφάσισε και μετά από σχετικές διαβουλεύσεις και εδώ με εσάς αλλά και με την Επιτροπή Προϋπολογισμών να μειώσει την εξάρτηση από εξωτερικές εταιρείες. Μειώσαμε τις συνολικά 133 συμβάσεις με εξωτερικούς συνεργάτες, εξωτερικές φίρμε, ε, συμβούλων κλπ. και θα τους αντικαταστήσουμε με 60 οργανικές θέσεις υπαλλήλων. ώστε να μειωθεί η εξάρτηση αυτή. Οι 60 αυτές θέσεις δεν έχουν καλυφθεί ακόμη, η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί. Η αντικειμενική αξιολόγηση θα μπορέσει να γίνει όταν θα έχει γίνει στελέχωση αυτή. Πάντως προχωρούμε σε μια καλύτερη εξισορρόπηση μεταξύ εσωτερικών πόρων και εξωτερικών εταιριών. Ρωτήσατε και για το Ευρωπάλ. Εμείς μετακινήσαμε το σύστημα από την αρχική προσέγγιση, την αρχική τηλεοπτική προσέγγιση και προχωρούμε σε παραγωγή ταινιών βίντεο, τις οποίες διαθέτουμε και σε άλλους. Αποτέλεσμα, μείωση του κόστους από αρχικά 9 εκατομμύρια σε νομίζω 5 εκατομμύρια που θα έχουμε για τον προσχή προπολογισμό. Δηλαδή φτάσαμε σχεδόν στο μισό θα ασχοληθούμε βέβαια ακόμη δατικότερα με την χρήση των προϊόντων αυτών, βίντεο κλπ. Στο δε διοικητικό πρόγραμμα εργασιών για την επόμενη, το επόμενο μισό της νέας δηλαδή ε, κοινοβουλευτικής περίοδου 2014-2016 θα κάνουμε σχετικές προτάσεις στο προεδρείο Για το ερώτημα τώρα του κ. Μάρτιν, ως διοίκηση εμείς απαντήσαμε όλες τις ερωτήσεις που μας υποβάλατε επισήμως. Ξεχωρίσαμε βέβαια τις ερωτήσεις οι οποίες αναφέρονται στο δημοσιονομικό έτος που αναφερόμαστε τώρα, αλλά προσπαθήσαμε να απαντήσουμε σε όλες τις ερωτήσεις σας. Κύριε Μιούλτερ, εσείς θέσατε το ερώτημα για το ημικύκλιο, νομίζω απήντησα ήδη. Η κυρία Γκρέσλε επίσης αναφέρθηκε στο ημικύκλιο, νομίζω και εκεί έχει καλυφθεί για το ερώτημα του συνταξιοδοτικού ταμείου, το οποίο είναι ένα θέμα το, που το έχουμε εδώ και αρκετό καιρό. Πρόκειται για ανεξάρτητο όργανο, οργανισμό, το οποίο δεν διαχειριζόμαστε εμείς. Αναμένουμε ότι θα μπορέσει να λειτουργεί ακόμα για έναν αριθμό ετών. Όμως, την άνοιξη του 2009, όταν ενέκυψε το Προεδρείο στο θέμα αυτό, είχαμε ήδη διαπιστώσει ότι ως Κοινοβούλιο είμαστε υπεύθυνοι για ενδεχόμενο έλλειμμα, δηλαδή υποχρώσεις για την καταβολή συντάξεων των Ευρωβουλευτών πρέπει να καλύπτονται, δηλαδή αν καταλήξουμε σε μια κατάσταση όπου το Ταμείο δεν διαθέτει πλέον πόρους, θα πρέπει να αναλάβει το Κοινοβούλιο. Θα θυμάστε όμως ότι και οι απαιτήσει απέναντι στο Ταμείο μειώθηκαν. Το 2009 σημειώθηκαν και κάποιες δικαστικές διαδικασίες. Έως τώρα όλες οι δικαστικές διαδικασίες κατέληξαν στο ότι οι σχετικές προσαρμογές που έκανε το Προεδρείο και σε ό,τι αφορά την συνταξιδοτική ηλικία και την πρόορη καταβολή των ε, συντάξεων, εφάπαυση δηλαδή, έγιναν δεκτά από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Για την τελευταία σας ερώτηση για την ανάθεση σε βουλγαρική εταιρεία. Εδώ τα πράγματα έχουν ως εξής. Η εντολοδόχος κατέθεσε δήλωση ότι δεν υπάρχουν συγκρουόμενα συμφέροντα. Σωστά είπατε ότι αυτό εντάσσεται μέσα στη συνήθεια διαδικασία. Και όντως έγινε στην προκειμένη περίπτωση. Ο εντολοδόχος όμως δεν είναι η βελγική διεύθυνση, αλλά η φύρμα στην Βουλγαρία. Είπατε ότι έχετε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με την βελγική εταιρεία. Όμως αντισυμβαλόμενος δικός μας είναι η βουλγαρική εταιρεία και η διαδικασία διεξάγεται σύμφωνα με τους συνήθεις κανόνες μας. Έχουμε δήλωση από την εντολοδόχο μας ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Τώρα, η κυρία Αγιάλα Σέντερ έθεσε ερωτήσεις σχετικά με την εσωτερικοποίηση καθώς και την επιστημονική υπηρεσία. Για το πρώτο θέμα, ιδίω όσον αφορά την ασφάλεια και αν κατάλαβα καλά ε, αναφέρεστε και σε αυτό και στην ασφάλεια δηλαδή μέχρι τώρα τα πράγματα κινούνται σύμφωνα με το σχεδιασμό. Ελπίζουμε ότι τελικά οι πληρωμές θα είναι χαμηλότερες, πάντως σίγουρα όχι παραπάνω. Έχουμε έμπιστους συνεργάτες οι οποίοι είναι πιστοί στο όργανο διότι είναι συμβασιούχοι μακρού χρόνου μπορούμε να του εκπαιδεύσουμε καλύτερα από συμβασιούχου ε, πολύ περιορισμένου χρόνου. Η δράση τους είναι πιο επαγγελματική και έχουμε και μία δομή με επαγγελματίες τμήματάρχες και διευθυντές, κάτι το οποίο αποτελεί σημαντική διαφορά για την διοίκηση των υπηρεσιών αυτών και αυτά μέσα σε μια βαθμιδόν διαδικασία η οποία κινείται όπως είπα βήμα-βήμα. Στον τομέα τώρα της πληροφορικής σημειώνονται ορισμένα προβλήματα σε ό,τι αφορά την πρόσληψη στελεχών. Όχι μόνο στον τομέα της πληροφορικής, σε πολλούς τομείς όπου χρειάζονται ειδικοί τεχνικοί εμπειρογνώμονες και για την πληροφορική και το ίδιο ισχύει για αρχιτέκτονες εφόσον απαιτούνται πρόσωπα που να έχουν εμπειρία με περίπλοκα έργα. Το ίδιο ισχύει και σε ορισμένες περιπτώσεις για διερμηνείς, εφόσον χρειάζονται πρόσωπα με, τις, με τους συγκεκριμένους γλωσσικούς συνδυασμούς που να μπορούν να εργάζονται ε, σε πλήονες γλώσσες. Άρα σε ε, πολλές τεχνικές, τεχνικού χαρακτήρα υπηρεσίες, υπηρεσίες έχουμε πρόβλημα με την πρόσληψη σε επίπεδο AD5 που επιβάλλει η μεταρρύθμιση Κίνοκ. Δεν έχουμε τις ίδιες δυσκολίες σε άλλους τομείς, για παράδειγμα ε, πολιτικών συμβούλων. Έχουμε όμως σημαντικό πρόβλημα, όπως είπα, για τεχνικούς εμπειρογνώμονες, πληροφορική κλπ. Και γι' αυτό δεν έχουμε μπορέσει να προσλάβουμε ακόμη τον αριθμό των 60 συνεργατών που θεωρητικά μπορούμε να προσλάβουμε. Το πρόβλημα αν, αν ευθύνεται σε αυτό η έψο, ο ενιαίος οργανισμός δηλαδή, δεν μπορώ να το απαντήσω το ερώτημα αυτό, δικαιολογείται όμως κανείς να το θέσει. Τώρα, για την ασφάλεια των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Όντως υπήρξαν ορισμένα συμβάντα, τα οποία οφείλονται κυρίως στο ότι το μη ασφαλές μέρος πρόσβαση στις υπηρεσίες μας. Ότι εκεί μπόρεσαν κάποιοι να σπάσουν κωδικούς. Το Προεδρείο ενέκυψε στο θέμα και σε βάθος αλλά και ταχύτατα και ενέκρινε τρία βήματα. Πρώτο, για τους επισκέπτες. Υπάρχει πρόσβαση στο Wi-Fi, πρόσβαση όμως η οποία επιτρέπει μόνο την πρόσβαση στο διαδίκτυο όχι σε εφαρμογές του Κοινοβουλίου. Ένα από τα προβλήματα που σημειώθηκαν ήταν ότι και απασχολούμενοι αλλά και ευρωβουλευτές χρησιμοποιούσαν το μη ασφαλές μέρος του διαδικτύου για να περνούν σε εφαρμογές του Κοινοβουλίου. Αυτή όμως η μη ασφαλής πρόσβαση δεν είχε το στόχο αυτό. Η μη ασφαλής πρόσβαση είναι για εξυπηρέτηση επισκεπτών και κυρίως επισκεπτών της μιας μέρας. Εξασφαλίζεται τώρα ότι οι επισκέπτες θα έχουν την πρόσβαση στο Wi-Fi, αλλά μόνο για χρήση διαδικτύου. Εφόσον τώρα εργαζόμενοι, υπάλληλοι δηλαδή ευρωβουλευτές ή άλλοι επιθυμούν πρόσβαση σε άλλες εφαρμογές του Κοινοβουλίου, τότε αυτό γίνεται μόνο μέσω πιστοποίησης, πιστοποιημένης δηλαδή πρόσβασης, δηλαδή κανείς είναι πιστοποιημένος χρήστης και μόνο με την έννοια αυτή μπορεί να έχει πρόσβαση στις σχετικές υπηρεσίες. Γνωρίζουμε όμως ότι πρόκειται για πιστοποιημένο χρήστη, ο οποίος έχει όντως το δικαίωμα πρόσβασης στις σχετικές ε, εφαρμογές και αυτό βεβαίως με τη σχετική τεχνολογία ασφάλειας. Τώρα, το τρίτο βήμα που ενέκρινε το Προεδρείο και που ελπίζουμε ότι θα μπορέσει να υλοποιηθεί μέχρι το καλοκαίρι, χρειάζεται μετάβαση σε ένα σύστημα που λέγεται Mobile Device Management, όπου θα γνωρίζουμε ακριβώς ποιος είναι ο χρήστης, τι είδους πιστοποίηση διαθέτει και τι είδους λογισμικό διαθέτει στο μηχάνημά του το οποίο να μην θέτει σε κίνδυνο είτε τον ίδιο το χρήστη είτε άλλους. Σύστημα το οποίο ήδη εφαρμόζεται στο Συμβούλιο βρίσκεται υπό μελέτη για εφαρμογή στην Κομισιόν και θα το εφαρμόσουμε και εμείς. Μια πολιτική δηλαδή που θα λέει ότι μπορώ να χρησιμοποιήσω η αδίποτε συσκευή, μπορώ να έχω η αδίποτε πρόσβαση και μπορώ να χρησιμοποιήσω η λογισμικό, η πολιτική αυτή δεν συμβιβάζεται με οποιαδήποτε έννοια ασφάλειας. Αυτό λοιπόν πρέπει να το έχουμε σαφώς υπόψη μας και γι' αυτό χρειάζονται Χρειάζονται μάλλον κάποιες αλλαγές, αλλαγές οι οποίες θα έχουν ως στόχο την προστασία των χρηστών, βεβαίως δεν μπορούν να τους προστατεύσουν απέναντι σε επιθέσεις που υποστηρίζονται από κράτη ή άλλα, άλλες τέτοιες οντότητες. Άρα δηλαδή αυξάνουμε το επίπεδο ασφαλείας απέναντι σε παρεμβάσεις ατόμων, πέραν αυτού όμως απέναντι σε κάποια μεγάλη οργάνωση ή κράτος, εκεί δεν μπορούμε να προσφέρουμε εγγύσεις. Και τελευταίο σχόλιο τώρα για την ε, κοινοβουλευτική υπηρεσία ερευνών. Αυτή έχει αρχίσει να λειτουργεί από 1η Νοεμβρίου. Βρέθηκα και την προηγούμενη εβδομάδα σε συνάντηση των συνεργατών όπου συζήτησαν τα θέματα τους η βιβλιοθήκη παραμένει ως ξεχωριστή διεύθυνση, υπάρχει όμως και μια πρόσθετη διεύθυνση, εκτός από την follow-up, που λέγεται Members Research Service, που έχει ως στόχο να καλύψει τα κενά τα οποία έχουμε εντοπίσει, ότι δηλαδή οι βουλευτές που συμμετέχουν σε μια κοινοβουλευτική επιτροπή υποστηρίζονται βεβαίως θαυμάσια από τη γραμματεία της Επιτροπής αλλά και από το Policy Department αλλά για κάθε θέμα είναι σωστό ότι υπάρχει και ένα 90% των βουλευτών που δεν είναι μέλη της Επιτροπής. Αυτό το 90% των βουλευτών όμως οφείλουν και αυτοί εν τέλει να λάβουν κάποιες ευθύνες διότι ψηφίζουν στην Ολομέλεια, διότι οφείλουν να βγουν έξω και να εξηγήσουν τους πολίτες τι συμβαίνει. Άρα χρειαζόμαστε εκτός από τις προφορίες για τα μέλη της συγκεκριμένη επιτροπής που τους χορηγούνται από γραμματείες και policy department, χρειαζόμαστε και πληροφορίες για το υπόλοιπο 90% των βουλευτών που δεν είναι ειδικοί, που δεν συμμετέχουν στη συγκεκριμένη επιτροπή, που ωστόσο έχουν κάποιο καθήκον να εκτελέσουν και άρα χρειάζονται πρόσθετες προφορίες. Ευχαριστώ. Ο πρόεδρος Τόιρερ, ευχαριστώ. Ο κύριος Μάρτιν ζήτησε ξανά τον λόγο και επισημένω εν προκειμένου ότι ο εισηγητής απεφάσισε ποιες ερωτήσεις θα υποβληθούν στο Γενικό Γραμματέα ή στο Κοινοβούλιο γενικότερα και ότι το Προεδρείο το έχει ενημερώσει ήδη ο κύριος Μάρτιν. Ευχαριστώ, θα είμαι σύντομος. Όχι κύριε Γενικέ Γραμματεύ, δεν συμφωνώ. Απαντήθηκαν τμήματα ερωτήσεων που σας υπέβαλε ο εισηγητής. Το ίδιο τώρα. Απαντήσατε σε πολλές ερωτήσεις τώρα που προέκυψαν από τη συζήτηση. Εγώ σας ανέπτυξα τα θέματα που με απασχολούν και θα το επαναλάβω. Μπορείτε πολύ εύκολα να μου απαντήσετε. Τώρα για την ασφάλεια στο διαδίκτυο γνωρίζετε εν τέλει ποιος κρύβεται πίσω από αυτές τις επιθέσεις. Ποια άτομα δηλαδή πιο συγκεκριμένα και μάλιστα ακούγεται και όνομα Ευρωβουλευτού. Ευχαριστώ κυρία Γκρέσλε. Ευχαριστώ για τις ε, πληροφορίες και τις διευκρινήσεις. Αντιλαμβάνομαι ότι στην υπόθεση αυτή της βουλγαρικής φύρμας Στάνισεφ δεν βλέπετε σύγκρουση συμφερόντων. Ναι, αλλά πώς ορίζεται τη σύγκρουση συμφερόντων. Εγώ πιστεύω ότι η υπόθεση αυτή χρειάζεται κάποια αντίδραση από μέρους μας. Είναι και ζήτημα αξιοπιστίας εν τέλει των ευρωπαϊκών θεσμών. Επίσης θα ήθελα να έχουμε κάποιες πληροφορίες σχετικά με αυτό το σώμα επιλογών έτσι, που προέβησε αυτή την ε, ανάθεση, επιλογή και ανάθεση. Δεν έχω άλλους εγγεγραμμένους. Σεις κύριε Γενική Γραμματεύ. επαναλαμβάνω προς τον κύριο Μάρτιν. Απαντήσαμε γραπτός στις ερωτήσεις που λάβαμε επισήμως. Δεν προέβημε σε επιλογή ποιον ερωτήσεων θα απαντήσουμε και ποιον όχι. Οι ερωτήσεις που μας υποβλήθηκαν επίσης και που δεν αφορούν το 2012, που θα μπορούσε κανείς να πει, κοιτάξτε δεν εντάσσονται μέσα στη διαδικασία απαλλαγής, δεν θα απαντήσουμε. Ωστόσο παρόλα αυτά αποφασίσαμε να απαντήσουμε. Βεβαίω δεν μπορούμε να απαντήσουμε παρά μόνο στι ερωτήσει οι οποίε εν τέλει μα διαβιβάζονται από την Επιτροπή. Ναι, θα απαντήσετε ναι ή όχι. Κατάλαβα τι είπατε κύριε Μάρτιν, είπατε ότι έχετε θέσει ορισμένε πρόσθετε ερωτήσει και θα τι εξετάσουμε. Επιμένω όμω ότι δεν μπορούμε να απαντήσουμε γραπτώς παρά μόνο τι ερωτήσει οι οποίε μα έχουν υποβληθεί γραπτό. Δεύτερο, για το θέμα της ασφαλείας. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι οι πληροφορίες αυτές προέρχονται από πολύ κοντά. Δηλαδή οι κωδικοί αυτοί άνοιξαν από κάπου πολύ κοντά. Δηλαδή από κάποιον ο οποίος χρησιμοποίησε μια δική μας διεύθυνση και που βρίσκεται στο άμεσο περιβάλλον του θυγωμένου προσώπου. Και όταν μιλώ για πάρα πολύ κοντά, μιλώ για το πολύ 50 μέτρα. Για το πολύ 50 μέτρα απόσταση από το θυγόμενο πρόσωπο. Αυτό μας εξήγησαν τουλάχιστον οι εμπειρογνώμονές μας. Άρα δεν προέρχεται από κάπου οπουδήποτε, αλλά από άμεση γυτνίαση, επαναλαμβάνω, το πολύ πέντε δεκάδων μέτρων. Δεύτερο, τώρα για την ερώτηση της κυρίας Γκρέσλε. Δεν προέβηνε σε αξιολόγηση για το αν πρόκειται σύγκρουση συμφερόντων ή όχι. Αυτό που είπα είναι ότι ο ή ανάδοχος κατέθεσε δήλωση ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα εξετάσουμε εγκύτερα, αλλά τυπικά τουλάχιστον είναι εντάξει. Έχει κατατεθεί δήλωση ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων όπως απαιτεί η διαδικασία. Και πέρασε από τα συνήθη όργανα, δεν επρόκειτο για μια μοναδική υποβολή προσφοράς, υπήρχαν νομίζω συνολικά 45 υποβολές προσφορών και η σχετική ε, αυτή η ε, υποβολή προσφορά βρισκόταν περίπου στο μέσον αυτό. Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστώ λέει ο πρόεδρος Δεν υπάρχουν άλλοι που ζητούν τον λόγο. Ρωτώ εάν το ελεγκτικό συνέδριο θέλει να προσθέσει κάτι. Thank Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Εν κατακλείδη, θα ήθελα να τονίσω ότι ε, το ελεκτικό συνέδριο συνιστά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να καταφέρει να πετύχει τον απαραίτητο συντονισμό να αφορά τη διαδικασία συμβάσεων προμηθειών μέσω μιας καλύτερης ε, καθοδήγησης. Αυτή είναι, αν θέλετε, η σημαντικότερη σύσταση που κάνουμε προς το Κοινοβούλιο για το τρέχον έτος. Ευχαριστώ και υπήρχε και μια ερώτηση της κυρίας Ορτής Βιλέγια προς τον εσωτερικό ελεγκτή, κύριο Κάλβιν. Μπορείτε να απαντήσετε στην ερώτηση της συναδέλφου. Ε, μπορείτε εδώ ή προτιμάτε γραπτός. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Μπορώ να απαντήσω τώρα. Επιβεβαιώνω ότι το σχέδιο δράσης το οποίο απορρέει από την εξωτερική αξιολόγηση του 2011 όντως ολοκληρώθηκε και το υπάρχουν απλώς κάποια επιμέρους στοιχεία για τα οποία χρειάζεται μια εξωτερική αδειοδότηση με ορίζοντα το 2020, δηλαδή αναθεωρημένος χάρτης συμπεριφοράς και δράσης για τον εσωτερικό ελεγκτή και θα ακολουθούμε εδώ πέρα κάποια συγκεκριμένα επαγγελματικά πρότυπα. Περιμένουμε τελική έγκριση από το Προεδρείο σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και πάλι, ο επιθυμεί να λάβει το λόγο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω απλώς τον Γενικό Γραμματέα για τις απαντήσεις που μας έδωσε και να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους για την συζήτηση που είχαμε και σας διαβεβαιώ ότι θα κάνω κάθε τι το δυνατό προκειμένου να συμπεριλάβω στο σχέδιο εκθεσή μου τα περισσότερα πράγματα τα οποία θίξαμε σήμερα. Στις 18 Φεβρουαρίου θα είναι διαθέσιμη και η εκθεσή μου. Σας ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά. Ο πρόεδρος Τόιρερ, ευχαριστώ. Τον εισηγητή, τον Γενικό Γραμματέα, τους εκπροσώπους του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τον Εσωτερικό Ελεγκτή, εδώ, αν δεν κάνω λάθος, λίγη η σημερινή ημερήσια διάταξη και μάλιστα και λίγο πριν από την ώρα που προβλεπόταν. Εδώ κλείνω την σημερινή συνεδρίαση. Αύριο ακρόαση για το λαθρεμπόριο τσιγάρων. Μετά η απογευματινή συνεδρίαση. Εμείς χρησιμοποιούμε όχι μόνο τη Δευτέρα και την Πέμπτη, αλλά από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη για να συνεδριάζουμε.